Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τους ε, συναδέλφους βουλευτές. Και επίσης να καλωσορίσω και τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να χαιρετήσω τον Ιβάιλο Κάλφιν, τον πρώην συνάδελφο, που δετέλεσε ευρωβουλευτής και μάλιστα σε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα υψηλού επίπεδου ε, υπό την προεδρία του Μάριο Μόντι. Θα ήθελα να καλωσορίσω εγκάρδια και τον Επίτροπο, τον κύριο Γκίντερ Έτιγκερ, που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλή. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε και αγαπητοί συνάδελφοι που λαμβάνετε μέρος σε αυτή την συνεδρίαση που θα επικεντρωθεί στη συνέχεια που θα πρέπει να δώσουμε στις συστάσεις που υπέβαλε η ομάδα υψηλού επίπεδου ε, για τους ιδίους πόρους. Μάλιστα την έκθεση ε, την παρουσίασαν πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 12 Ιανουαρίου. Και σήμερα έχουμε την ε, δυνατότητα, την ευκαιρία και την τύχη θα έλεγα να συζητήσουμε αυτό το θέμα παρουσία των βουλευτών από τα κοινοβούλια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή, η έκθεση υψηλού επίπεδου, ήταν το επιστέγασμα εκτενών διαβουλεύσεων και μια διάσκεψη με θέμα τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού που έγινε στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου του 2016. Για τα διαδικαστικά να σας υπενθυμίσω δύο-τρία πράγματα. Καταρχήν θα ακούσουμε τους καλεσμένους μας τον Επίτροπο, τον Αλάλα Μασούρ, που επίσης ε, ήταν μέλος της ομάδας υψηλοεπέδου, θα έρθει όμως αργότερα στις 10. Θα ακούσουμε τον Ιβάιλο Κάλφιν και δύο πανεπιστημιακούς, την κυρία Κώστας Άλντολφ και την κυρία Ντανούσα Νερούντοβα. Έχετε μάλιστα και δελτία που μπορείτε να τα συμπληρώσετε με το όνομά σας και το κοινοβούλιο από το οποίο προέρχεστε για να λάβετε το λόγο. Κανονικά θα έχει τρία λεπτά χρόνο ο καθένας. Αν ο κατάλογος ομιλητών είναι εκτενής, ίσως περιοριστούμε στο δίλεπτο. Θα φροντίσω να δίνω το λόγο σε δύο βουλευτές και σε έναν ευρωβουλευτή. Αυτά ως προς το διοργάνωση της πρωινής αυτής συνεδρίασης. Πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στον Επίτροπό μας, τον κύριο Γκίντερ Έτιγκερ, που μέσα σε 15 περίπου λεπτά θα μας κάνει μια εισαγωγή. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Verehrter Herr Vorsitzender, Αξιότιμε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να παρουσιάσω σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων να παρουσιάσω κάποιες ε, απόψεις μας για το θέμα των ιδίων πόρων για το θέμα των εσόδων των μελλοντικών κοινοβουλίων. Και αυτά θα τα πράξω με βάση την έκθεση του κυρίου Μάριο Μόντι, ο οποίος ε, από κοινού με άλλες ε, εξέχουσες προσωπικότητες, τις οποίες ε, διόρισε το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, ανά τρεις διορίστηκαν αυτοί. Στο τέλος του έτους λοιπόν ο κύριος Μάριο Μόντι παρουσίασε την έκθεσή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Λαμασούρ και τον κύριο Κάλφιν για το γεγονός ότι με την εμπειρία τους, ε, την εμπειρία την οποία συνέλεξαν όλες αυτές τις ε, δεκαετίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι δύο συνέβαλαν τα μάλα στις εργασίες μας και σήμερα έχουμε και τη χαρά και την τιμή να τους έχουμε κοντά μας ως εισηγητές. Η έκθεση λοιπόν αναφέρεται σε μία εντολή που δόθηκε το Δεκέμβρη του 2013. Τότε λοιπόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε ε, αρμόδιος ήταν ο συνάδελφός μου ο κ. Λεβαντόφσκι. Τότε λοιπόν προτάθηκε ένας προϋπολογισμός 7 ετών ο οποίος εγκρίθηκε την τελευταία στιγμή και ο οποίος προϋπολογισμός περιλάμβανε διαφόρων ειδών μέτρα και επίσης ε, περιλάμβανε και την εντολή από το Κοινοβούλιο, το ε, Συμβούλιο και την Κομισιόν προς τον κύριο Μόντι και την ομάδα του να ε, καταθέσουν τη σχετική εισήγηση. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος ότι η έκθεση που έχουμε μπροστά μας εγκρίθηκε ομόφωνα. Αυτή η ομοφωνία, το γεγονός ότι συμφωνούν και τα δέκα μέλη της Επιτροπής αποτελεί η ομοφωνία τη βάση για να μπορούμε να εξάγουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη οι προτάσεις ε, που περιλαμβάνονται ε, θα πρέπει να οδηγήσουν στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που σας προτείνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση δικές μου προτάσεις ή κομισιόν εφέτος θα ξεκινήσει τις ε, εργασίες για το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο πριν από το τέλος του 2017 υπάρχει η δέσμευση να υποβληθεί το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020. Αυτό το πλαίσιο ε, να παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο. Τα πράγματα όμως δεν θα είναι απλά, γιατί ζούμε σε μια ταραγμένη εποχή και ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιε θα είναι οι προτεραιότητε το 2020, το 2026. Θα είναι τότε σημαντικό το προσφυγικό, η ανεργία των νέων, η προστασία των συνόρων. Ποια θα είναι τα φλέγοντα θέματα. Θα είναι ε, απαραίτητο να γίνονται επενδύσεις ε, στην καινοτομία και ε, στην υποδομή έτσι ώστε η Ευρώπη να καθίσταται ανταγωνιστική. Αυτά είναι απρόβλεπτοι παράγοντες και αυτό που επίσης επιτείνει την ε, ανασφάλεια είναι το Brexit και οι επιπτώσεις που θα έχει στη δημοσιονομική μας πολιτική. Γιατί μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Αυτό που είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η έκθεση Μόντι περιλαμβάνει μία σειρά προτάσεων για τη διαμόρφωση των εσόδων χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρξει αλλαγή στη συνθήκη ή στις συνθήκες. Οι προτάσεις δηλαδή κατατίθενται με βάση την ε, εφαρμογή του πρωτογενούς δικαίου. Και αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι καμία πρόταση δεν μπορεί να βασίζεται σε χρέος στην ανάληψη χρέους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δεν θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα που θα μας οδηγεί στις ε, τράπεζες. Όχι, κάθε άλλο, θα πρέπει να επικρατήσει η αρχή ότι η Ευρώπη θα δύναται να δαπανά τα χρήματα που εισπράττει. Και αυτό σε αιτήσια βάση. Το ευρωπαϊκό λοιπόν επίπεδο παραμένει το μόνο επίπεδο το οποίο ε, θα ξεκινήσει τη μελλοντική του πορεία, το ευρωπαϊκό αυτό επίπεδο, χωρίς χρέη. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι η έκθεση Μόντι δεν αποβλέπει σε αυτόματα έσοδα. Δηλαδή πρόκειται κατ' ουσίαν για μία αναδιάταξη, αναδιάταξη των εσόδων η οποία αναδιάταξη αυτή θα πρέπει και στο μέλλον να λαμβάνεται καθοριστικά υπόψη. Κατά πόσον θα μιλάμε στο μέλλον για το 1% του ΑΕΠ όχι, αυτό παραμένει μια ανεξάρτητη απόφαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η έκθεση Μόντι δεν καθορίζει το ανώτατο όριο των εσόδων, απλά προβλέπει εργαλεία για το πώς ακριβώς ε, θα υπάρχει κάποια ισορροπία στα προτινόμενα έσοδα. Επίσης, η έκθεση Μόντι καθορίζει και μία πορεία και λέει καταργούνται οι εκπτώσεις. Καμία έκπτωση πλέον. Ε, στο πλαίσιο του νέου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και ε, κάτω από το πρίσμα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσουν οι Βρετανοί, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες ε, έχουν διεκδικήσει και αποκτήσει ουσιαστικές εκπτώσεις, παρότι οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι καθαρή συνεισφορής τώρα πλέον έχει φτάσει η στιγμή να μην υπάρχει πλέον καμία εξαίρεση από τις αρχές που διέπουν τα έσοδα και ως εκ τούτου το θέμα της ε, χρηματοδότησης των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι όποιος επιθυμεί να παρατείνει χορήγηση και αναγνώριση εκπτώσεων ή επιθυμεί να έχει κάποιες εκτός ορισμένα θέματα, πρέπει να το αιτιολογεί. Ως εκ τούτου, κατά την επόμενη δεκαετία δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχουν εκπτώσεις, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, τα έσοδα θα πρέπει να βασίζονται σε ε, αναγνωρισμένες διαδικασίες. Όλοι οι μηχανισμοί διόρθωσης θα πρέπει να καταργηθούν. Αυτά αναφέρει η έκθεση Μόντι. Αν δούμε, αν λοιπόν λιγάκι την δημοσιονομική δομή των τελευταίων ετών, θα διαπιστώσουμε ότι στην αρχή βασιστήκαμε κατά κύριο λόγο στους δασμούς. Οι δασμοί ήταν εκείνοι που χρηματοδοτούσαν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και με την πάρδα των ετών, με τις ε, συμφωνίες που συνήφθησαν, ΣΕΤΑ, οι διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία, με την Νέα Ζηλανδία, ακόμα και στη συμφωνία TTIP, αλλά και σε κάθε συμφωνία με κάθε χώρα που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου δεν ήταν πλέον εμπορικός εταίρος αλλά μέλος της κοινή αγοράς, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κατέπεσαν οι δασμοί. Ως εκ τούτου, οι δασμοί δεν μπορεί να είναι πλέον η σταθερή βάση για να προκύπτουν έσοδα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα Παραδείγματο χάρη αυτό που επιβλήθηκε στη Microsoft ή και σε άλλες εταιρείες, τέτοιου είδους πρόστιμα παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου οι κυρώσει και αυτές δεν είναι σταθερή πηγή εσόδων. Ε, αν μια περίπτωση, παραδείγματο χάρη, να υποθέσουμε, μα αποδίδει 11 δισεκατομμύρια ευρώ, μα αυτή είναι μια έκτακτη πηγή εσόδου, η οποία βέβαια χρησιμοποιείται και για συμψηφισμό και η οποία πηγή αυτή δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ε, και να εγγράφεται, ως σταθερή πηγή εσόδου και να εγγράφεται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το τρίτον, ε, τα ποσοστά του φόρου κύκλου εργασιών είναι τόσο περίπλοκα έτσι ώστε κανείς πλέον δεν κατανοεί το τι ακριβώς ε, επιβάλλουν τα κράτη-μέλη και με βάση ποια φόρμουλα. Ε, το να απλουστευτεί λοιπόν ο υπολογισμός του φόρου κύκλου εργασιών, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα καθήκον μας. Και όσον αφορά τη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αυτό που παίζει ρόλο είναι κατά πόσον είναι καθής, κανείς ε, καθαρός συνεισφορέας ή κατά πόσον είναι χρήστης αυτών των προϋπολογισμών. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ε, διάφορες ε, ε, διάφορους ε, υπολογισμούς. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι ένας καθαρός συνεισφορέας, που είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκα εγώ, ένας καθαρός ε, συνεισφορέας, ναι πράγματι είναι η Γερμανία, αλλά σε γενικές γραμμές εποφελείται πλήρως από ευρωπαϊκά προγράμματα. Από ένα ευρώ το οποίο καταβάλλεται από τη δική μου την πόλη τη Γερμανία στην, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ο οποίος, ε, ε, το οποίο αυτό διατίθεται για διαρθρωτικά ή οποιαδήποτε άλλα προγράμματα, ας μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε εταιρείε ε, την Hochtief και πάρα πολλές άλλες εταιρείε οικοδόμησης και ανάληψης έργων, το 40% επιστρέφει. Άρα δηλαδή μπορεί κανείς ε, να θεωρήσει ότι ο καθαρός συνεισφορέας είναι και εκείνος ο οποίος επωφελείται πλήρως στον, πλήρη, ε, στον τελικό απολογισμό. Για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες δομές εσόδων. Επίσης, να σας πω, εμείς είμαστε ευγνώμονες για το ότι η Επιτροπή Μοντή έχει ε, εξετάσει όχι μόνο τα έσοδα, αλλά και τα έξοδα. Και είναι ιδιαίτερα αυστηρή και στο θέμα των εξόδων. Και τίθεται το βασικό ερώτημα κατά πόσον προκύπτει υπεραξία. Αν προκύπτει υπεραξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά πόσον προκύπτει υπεραξία και για εθνικές πολιτικές, ε, δηλαδή ε, αν τελικά προκύψουν νέα εργαλεία για τους ίδιους πόρους, κατά πόσον αυτά θα βοηθήσουν στη συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μιλάμε δηλαδή για υπεραξία που προκύπτει από δαπάνες που ε, έχουν εγκριθεί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μιλάω ξεκάθαρα για δαπάνες για εκταμείευση κοντιλίων. Γι' αυτό λοιπόν η προστασία των συνόρων, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική προληπτική, το προσφυγικό, η αντιμετώπιση του μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, προφανώς αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και άλλοι τομείς όπως παραδείγματος χάρη η ευρωπαϊκή έρευνα. Αυτά για την εκταμείευση κονδυλίων και τις δαπάνες. Όσον αφορά τα έσοδα, θα πρέπει να προβάλλουμε αυτό που ε, έχει αναφέρει ο κύριος Λαμασούρ, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν συνέργειες ε, που να καθορίζουν τις εθνικές πολιτικές. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η Επιτροπή Μόντι έχει στα χέρια της νέα εργαλεία για νέες πηγές εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις. Όλα αυτά, κατά κάποιον τρόπο, είναι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής. Έχουμε λοιπόν δύο μεγάλα μπλοκ, τα οποία θέλω και να σας αναφέρω. Το ένα μπλοκ είναι η περιβαλλοντική πολιτική, προστασία του κλίματος, ε, αποδοτική χρήση της ενέργειας, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν ήταν δυνατόν τους ε, ευρωπαϊκούς στόχους, την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα να τη δεσμεύσουμε σε ε, να την εντάξουμε σε ένα κομμάτι του συστήματος ε, ανταλλαγής εκπομπών. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα είχαμε συνδυασμό της, της πολιτικής μας με την ενεργειακή πολιτική. Ναι, αναφερθώ σε κάτι άλλο, ε, στον φόρο που θα επιβάλλεται στις διατραπεζικές συναλλαγές. Εάν λοιπόν περιοριστούν οι κίνδυνοι στον οικονομικό τομέα με τη συγχρηματοδότηση του προπολογισμού, θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να συνδυάσουμε την δημοσιονομική πολιτική με πολλέ άλλε πολιτικέ. Αυτό που μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, την Άνοιξη ε, θα έρθω εδώ πολλέ φορέ να σα επισκεφτώ. η δική μα φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι με το πακέτο για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 να καταθέσουμε ρεαλιστικές προτάσεις με βάση την πρόταση Μόντι. Ε, θα ήθελα να προτείνω στους ε, ευρωβουλευτές ε, από τα κράτη-μέλη αν θέλουν να έρθουν να με επισκεφτούν και μένα ή αν θέλετε και τους ε, συνεργάτες μου, αλλά και εμείς μπορούμε να σε επισκεφτούμε στο Παρίσι, στο Δουβλίνο, στη Βιέννη, στη Ρώμη, ε, να σε επισκεφτούμε οποτεδήποτε θα συνεδριάζουν οι αρμόδιες ε, επιτροπές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Μάλιστα. Ακούσατε τα χειροκροτήματα. Πολλά υποσχόμενα χειροκροτήματα. Είμαστε στο τέλος ενός κύκλου, σίγουρα. Και αυτός ο προπολογισμό ε, χαρακτηρίζεται από τη λιτότητα, αυτό, αυτή είναι η σφραγίδα του και είναι κάπως αναχρονιστικός στο βαθμό που διαμορφώθηκε ε, πριν από 7 χρόνια στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και είναι περισσότερο καθρέφτης αυτού που συνέβη στο παρελθόν παρά αυτού που θα συμβεί. Και όταν προκύπτει μια κρίση, φυσικά έχουμε ατελείωτες δυσκολίες να βρούμε τα μέσα για να τα αντιμετωπίσουμε. Μιλήσατε για τους ίδιους πόρους, για, τα, ε, για τους φορολογικούς δασμούς, για τους ε, δασμούς, όπως έχουμε όλο και περισσότερες ε, ε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Ε, όλο λοιπόν και συρρυκνώνονται τα, αυτά τα έσοδα, μόνο το 10% είναι. Και επίσης έχουμε και περίπλοκους μηχανισμούς εκτόσεων, που θα εξαφανιστούν βεβαίως μια και το 80% του προπολογισμού ξαναπηγαίνει στα κράτη-μέλη μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής ή, μέσω των, του Ταμείου Συνοχής, έχουμε αυτή την λογική της δίκαιης ε, επιστροφής και το κάθε κράτος α, μέλος ουσιαστικά υπολογίζει τι έδωσε και τι πήρε και ουσιαστικά θέλει να πάρει αυτά που έδωσε. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη, δεν είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι με βάση το πνεύμα της ε, Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, θα πρέπει να τα ξεφορτωθούμε. Η έκθεση Μόντι προφανώς είναι ένα έγγραφο το οποίο θα μας βοηθήσει όλους, ούτω ώστε να γίνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός η απεικόνηση της θέλησης για πρόοδο στην Ευρώπη. Κύριε Κάλφη, εσείς που συμμετείχατε σε αυτή την ομάδα εργασίας, θα θέλατε τώρα να μας ε, πείτε τις παρατηρήσεις σας και το όραμά σας. Πώς θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα προπολογισμό που θα μπορέσει να δείξει ότι έχει ένα δυναμικό και ότι δεν είναι εντελώς αδύναμη απέναντι στις κρίσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Αχτούς που έβαλε αυτό το θέμα ε, προσυζήτηση σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό και τον εθνικό και τον ευρωπαϊκό, μην ξεχνάμε ότι τα κοινοβούλια ε, αποφασίζουν πώς λέγονται τα χρήματα και πώς αναδιανέμονται, για ποιες πολιτικές, ποια είναι η αποτελεσματικότητα της διανομής ε, και ποιο είναι το αποτέλεσμα, όλων αυτών των προσπαθειών για τους πολίτες από αυτή την δημοσιονομική προσπάθεια. Επομένως, η συζήτηση για οποιαδήποτε αλλαγή στις, στα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναπόφευκτα ένα σημείο συζήτησης μεταξύ των εκλεγμένων εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων δηλαδή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τούτου λεχθέντος, να σας πω ευθύ εξ αρχής ότι αυτό που προτείνουμε στην έκθεση δεν είναι μια μάχη μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δεν είναι ε, ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη εξουσία ε, εμείς ή το εθνικό επίπεδο ή τα θεσμικά όργανα μεταξύ τους. Θέλουμε να εξορθολογήσουμε τη διαδικασία, γιατί χωρίς αυτή θα χάσουμε την αρχή της επικουρικότητας, που σημαίνει ότι εθνικά κοινοβούλια ε, σε οποιαδήποτε φάση θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν επί του ε, ευρωπαϊκού προπολογισμού και επί των εθνικών συνεισφορών και το πώς ξοδεύονται τα χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η πρόταση εξορθολογικεύει τη χρήση των δημοσίων οικονομικών χωρίς, και το επαναλαμβάνω και το τονίζω, μείωση της δυνατότητας παρέμβασης των εθνικών κοινοβουλίων και εθνικών κυβερνήσεων να παρέμβουν, να πούν την άποψή τους και μέσω διαδικασιών συνενετικών, ούτω ώστε να αποφασιστεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Έτιγκερ για την παρουσίασή του και για την διάθεσή του από την αρχή της προσπάθειας να λάβει υπόψη του τις προτάσεις που περιλάβαμε στην έκθεση αυτή της ομάδας υψηλού επίπεδου. Όπως μόλις σας είπε, το 2017 είναι η χρονιά όπου θα αποφασίσουμε για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μετά το 2020. Και φοβάμαι ότι δεν θα είναι η μόνη αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων όλων των διαδικασιών που είναι να εξελίξει και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιασδήποτε αλλαγές συμβούν και αν συμβούν στην Ένωση, ο προπολογισμό θα είναι σίγουρα ένας, ε, μία από αυτές τις αλλαγές. Επομένως τώρα είναι η στιγμή να σκεφτούμε πώς θέλουμε να τον βελτιώσουμε, πώς θέλουμε να βελτιώσουμε την όλη διαδικασία συλλογής και δαπάνης των δημοσίων του δημοσίου χρήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε διάφορα εργαλεία, θα ήθελα να το πω. Ε, έχουμε στον εθνικό προπολογισμό, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και διάφορους μηχανισμούς σταθερότητας, κυρίως στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά είναι υπό τη μορφή ε, ε, επιχορηγήσεων ή εγγύσεων για τα χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει λοιπόν τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά να διαμορφωθούν ε, μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο, σαν ένα πακέτο. Μεταρρύθμιση λοιπόν του ευρωπαϊκού προπολογισμού γιατί χρειάζεται. Είναι κάτι σπάνιο αυτό που θα σας πω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια και κατάληξαν σε μία έκθεση σχεδόν 100% συνενετική. Όλες αυτές οι αλλαγές που προτείνουμε είναι πραγματικά απαραίτητες εξού και συνένεση. Και υπάρχουν ελάχιστα επιχειρηματικά υπέρ του τρέχοντος ε, συστήματος, του να διονυστεί δηλαδή και στο μέλλον. Γιατί όμως. Γιατί το σύστημα αυτό δεν είναι ούτε διαφανές, ούτε κατανοητό. Κανένα στην Ευρώπη δεν μπορεί να εξηγήσει στους πολίτες γιατί μια δεδομένη χώρα πληρώνει τόσα λεφτά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Έχετε εκατοντάδε εξαιρέσει, ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο δέντρο, α πούμε, και μια ολόκληρη διαδικασία για να διαπραγματευτούμε την, ε, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η διαδικασία γίνεται αδιαφανώ μέσα στο Συμβούλιο και τελικά δεν υπάρχει καμία εξήγηση γιατί η χώρα Χ, πούμε, πληρώνει τα λεφτά ψή και αντιστοίχω δεν είναι εφικτό να ενημερώσουμε του φορολογούμενου γιατί πληρώνουν τόσα και να καταλάβουμε και τι παίρνουν σε αντάλλαγμα. Δεύτερον, βλέπουμε τώρα ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό επηρεάζεται από όλη τη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, διαμορφώνεται για 7 χρόνια υπομορφή εθνικών ποσών, δηλαδή ποσά που επιστρέφουν στα, στα κράτη-μέλη, αυτός ο προπολογισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες των πολιτών. Αυτή τη βδομάδα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν ε, στη Μάλτα το θέμα της μετανάστευσης. Και αυτό είναι από τα θέματα που σίγουρα είναι πολύ σημαντικά για όλους. Το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά μαζί αλλέγγυα στην πρόκληση της ε, μετανάστευσης. Και αυτό η αντίδραση εξαρτάται και από, την, ε, από τη δύναμη του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Είναι καλό παράδειγμα αυτό. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη που μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση της μετανάστευσης χωρίς τη βοήθεια των υπόλοιπων χωρών. Είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφέστατη προστιθέμενη αξία, όπου μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο δαπανών, που, λόγω των πολιτικών, και μπορεί να δώσει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιοδήποτε μεμονωμένο κράτο μέλο. Παράλληλα όμω, ε, αυτό ποτέ δεν ελήφθη υπόψη στον προπολογισμό τότε που Υιοθετήθηκε το 2012. Υπάρχει περιορισμένη ευελιξία. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε φέτο, τα επόμενα χρόνια κτλ. Αλλά είναι περιορισμένη και σίγουρα δεν είναι στο ύψο των προσδοκιών των πολιτών. Επομένω, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα προπολογισμό ο οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τι προκλήσει και τι ε, προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Φυσικά στην εκθεσή μα εστιάζουμε στα έσοδα Φυσικά γιατί αυτή ήταν η εντολή που λάβαμε από τα τρία θεσμικά όργανα. Για πρώτη φορά το Συμβούλιο μάλιστα συμφώνησε να δώσει μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα το, τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα των εσόδων και με το Κοινοβούλιο. Μέχρι τώρα όλες οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδείκνυαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μουγκό στο θέμα των ε, εσόδων του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και το απο... αποφάσισαν για τον προπολογισμό κυρίω ε, τα κράτη-μέλη και κυρίω οι, οι κυβερνήσει. Ελάχιστε χώρε είχαν ε, εντελεχή συζήτηση για το πώ ε, θα διαμορφωθεί η εθνική συνεισφορά πριν ε, υιοθετηθεί το εθνικό το μας πλαίσιο. Χωρίς λοιπόν το, τους ερετούς προσώπους, χωρίς τους κοινοβουλευτικούς αποφασιζόταν αυτά τα πράγματα. Εμείς λοιπόν προτείναμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, να ξεφορτωθούμε τι παραχωρήσεις, εξαιρέσεις, μειώσεις, εκτόσεις, επιστροφές κτλ κάτι που καθιστούσε τον προπολογισμό εντελώ ακατανόητο. Και χαοτικό. Και δεύτερον, θα πρέπει να αποκαλύπτουμε τις πηγές εσόδων και να αυξήσουμε τις πηγές χωρίς να φορολογήσουμε περισσότερο τους πολίτες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι τμήμα των ε, δημοσιονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξάλλου, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν προτείνουμε τι πηγέ. Ε, Επίση, το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων ε, να παίρνουν αποφάσεις ε, το κρατάμε. Δεν θέλουμε ευρωπαϊκού φόρου, δεν προτείνουμε τίποτα το οποίο θα διαμορφώνεται πίσω από την πλάτη των εθνικών κοινοβουλίων. Όλα όσα λέμε είναι, θα αποφασίζονται από κοινού, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια ούτως ώστε να βελτιωθεί ο προπολογισμό. Έχουμε συγκεκριμένε προτάσει για εναλλακτική χρηματοδότηση, εναλλακτικές πηγές. Ε, θέλουμε ε, να αυξήσουμε κατά 5% τους ίδιους πόρους τουλάχιστον. Ο Πίρπος και τώρα ανέφερε ότι θα αυξηθούν λιγότερο από 20% και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Δεν μιλάμε για φορολογία μόνο και μόνο για να δημιουργηθούν ποσά μιλάμε για έσοδα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι μπορεί να κάνει. Και όταν μιλάμε για κοινή φορολογική βάση, αυτό συνδέεται με την φοροαποφυγή. Όταν μιλάμε για περιβαλλοντικούς φόρους, όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά και αυτές που, εισάγουν τα... εξάγουν δηλαδή τα αγαθά τους σε εμάς, ε, όχι, θα πρέπει να ε, μην μπορούν να έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί αδιαφορούν εντελώς για το περιβάλλον. Αυτές, αυτοί οι πόροι ε, δημιουργούνται λόγω της ύπαρξης Ευρωπαϊκής Ένωση. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπήρχαν καν αυτές αυτές οι πηγές χρηματοδότησης. Να τελειώσω με δύο φράσεις για το τι εμείς προτείνουμε και το πώς βλέπουμε τώρα η διαδικασία στο μέλλον. Όπως είπα ήδη, δεν είναι δυνατόν να έχουμε αποτελέσματα τα εθνικά κοινοβούλια δεν συμμετέχουν στη διαδικασία και δεν συμφωνούν. Νομίζω ότι ο διάλογος δεν θα γίνεται μία φορά το εξάμεινο ή το, χρόνο, αλλά υπό τη μορφή ε, συζητήσεις σε group ή σε task force κτλ. Και θα είναι διαρκής και είναι σημαντικό. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί εσωτερικά και σε εθνικό επίπεδο επίση. Και σε περιφερειακό επίπεδο μερικές φορές, γιατί και οι περιφέρειες ε, προφανώς και ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τις αφορά. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τις αλλαγές που υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι θα αλλάξει. Όχι γιατί ένα από τα κράτη-μέλη θα φύγει τελικά από την Ένωση, αλλά γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι τα καθαρά, ας πούμε, έσοδα, τι, τι, τι, δίνεις και τι παίρνει, αλλά ποια είναι η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το να είσαι μέλος αυτής. Και ποια είναι τα εργαλεία του κάθε κράτους μέλους για να, συμμετέχουν, για να συμμετέχει. Ε, αυτό το θέμα λοιπόν ε, θα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο, ε, με, ίσως με μια εργαλειοθήκη ε, που θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε αυτή την αξία. Ευχαριστώ. Je remercie. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην συνάδελφο Ιβο Κάλβιν, Ιβάιλο Κάλβιν, για την ε, σύνοψη της έκθεσης, για την ανάλυση και τις συστάσεις της ομάδας αυτής υψηλού επίπεδου υπό την Προεδρία του Μάριο Μόντι. Και διαπιστώνω ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ ελπιδοφόρα, πολλά υποσχόμενα. Και στην Επιτροπή Προπολογισμών, επειδή πιστεύουμε ότι καθήκον μας είναι να υποβάλουμε έναν ε, κατανοητό και βανάγνωστο για τους Ευρωπαίους πολίτες προϋπολογισμό, να κάνουμε το καθήκον μας για να έχει κάποια απήχηση η Ευρώπη στους Ευρωπαίους. Καταλήξαμε λοιπόν σε αυτό το πίνακα που έχει και η έκθεση της ομάδας εργασίας όταν αντιμετωπίζουμε μια κρίση, όταν δεν έχουμε τα μέσα να την διορθώσουμε, ουσιαστικά έχουμε trust funds, κάποια καταπιστεύματα, κάποιου δημοσιονομικού δορυφόρου για την Αφρική, για τη Συρία, δημοσιονομική ικανότητα για την Τουρκία, κάποια χρηματοδοτικά μέσα που είναι τόσο δυσανάγνωστα, τόσο κατανόητα. Και μάλιστα εδώ απευθύνομαι στους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εσείς Πώς ελέγχεται τις συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα διάφορα θεσμικά όργανα. Πώς γίνεται η κοινοβουλευτική συζήτηση. Δεν έχει έρθει ακόμη ο Αλένα Μασούρ. Καταφθάνει, καταφθάνει. Καλώς ήρθατε κύριε Λαμασούρ. Ο Αλένα Μασούρ συμμετείχε και αυτό στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Επίτροπο Ότιγκερ που φαίνεται πραγματικά αποφασισμένος να οδηγήσει τον προϋπολογισμό στην ίδια κατεύθυνση με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου. Μας ανέλησε την πρόταση, επέμεινε στην ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και στην βούληση να ανέλθει το ποσοστό των ιδίων πόρων. Σήμερα είναι 15 δισεκατομμύρια από τα 158, 10% δηλαδή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι μόνο ιδίοι πόροι. Θέλει να αυξήσει αυτό το ποσοστό από τα 10% στα 50%. Σημαντική πρόκληση και μια ναι, και θα έχουμε ιδίου πλέον πόρου, δεν θα μιλούμε για τι δίκαιε πια επιστροφέ και όσο λιγότερο θα μιλούμε για τι ε, δίκαιε επιστροφέ, θα έχουμε περισσότερο ένα κοινό όραμα και όλο και μεγαλύτερη συμφωνία για αυτό το κοινό όραμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα είναι μασούρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σα ζητώ συγγνώμη που δεν ε, ήμουν παρόν από την ε, έναρξη των εργασιών σα. Αλλά είχα πρόβλημα με τι συγκοινωνίες. Χαίρομαι ιδιαίτερος για την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων με αυτούς που κατέχουν την ε, δημοσιονομική κυριαρχία, δηλαδή τους ε, βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, παρουσία του Επιτρόπου Έτιγκερ, για το θέμα αυτό που είναι η μαύρη τρύπα της ευρωπαϊκής πολιτικής συζήτησης. Σχεδόν σε καμία χώρα Κανένα, κανένα πολιτικό κόμμα, κανένα τουλάχιστον κυβερνών κόμμα, δεν τολμά να θίξει το ζήτημα του κοινοτικού προϋπολογισμού και της χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, πέραν αυτών που είπε ο Ιβάιλο Κάλφιν, και συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι τώρα, θα ήθελα να επιμείνω σε τρία σημεία. Πρώτον, οι προτάσεις της ομάδας υψηλού επίπεδου σέβονται απόλυτα τις συνθήκες το γράμμα και το πνεύμα των, ευρωπαϊκών συνθήκων γίνεται απολύτως σεβαστό. Και όχι μόνο σέβονται το γράμμα και το, το πνεύμα του νόμου, αλλά ακριβώς επανέρχονται στην πηγή των ευρωπαϊκών συνθήκων που προβλέπουν από την πρώτη μέρα λειτουργία τους, γιατί στις 25 Μαρτίου θα εορτάσουμε την 60η επέτειο της ε, Ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώμης. Προβλέπουν λοιπόν ότι οι δαπάνες που ε, προβλέπουν οι ευρωπαϊκές πολιτικέ χρηματοδοτούνται από ένα κοινοτικό προπολογισμό που έχει ιδίου πόρου, δηλαδή φορολογικού πόρου, φορολογικά έσοδα ε, που είναι τελωνιακοί δασμοί κυρίω και δρομολογούνται προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει το δικαίωμα ή την ικανότητα συλλογής φόρων, αλλά σε ένα πλαίσιο που καθορίζει ο φορολογικός κυρίαρχος, ο δημοσιονομικός κυρίαρχος που είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ένα ποσοστό ιδίων πόρων και ένα περιθώριο ελιγμών ως προς το ποσοστό αυτών των ιδίων πόρων. Όπως ε, ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη για τους ε, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς ε, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ίσως κάπως ως ιδιάζουσα τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να θεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, γεωγραφικά ε, υπερέχει, αλλά αυτή είναι, αυτός είναι ο παραλληλισμός. Δεύτερον, ίσως ε, το πιο εντυπωσιακό σημείο της έκθεσης είναι ο πίνακας που ε, κατέρτισε και η Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το στερέωμα, τον αστερισμό των δορυφορικών αυτών μέσων και των μικροπροϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πολλαπλασιάζονται στο περιθώριο του κοινοτικού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών. Και μια και ο κοινοτικό προπολογισμό είναι πολύ περιορισμένος και εδώ και 20 χρόνια έχει de facto ένα ανώτατο όριο το 1% του ΑΕΠ και ενώ από τις συνθήκες και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες και έχουν προσθεθεί νέες πολιτικές και απαιτούν μια ελάχιστη χρηματοδότηση, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια στον κοινοτικό προϋπολογισμό και γι' αυτό τα αναζητούμε αυτά τα κονδύλια αλλού. Ε, φτιάχνοντας μικροπροϋπολογισμούς με διάφορους τίτλους και ονόματα για να χρηματοδοτήσουμε κάποιες νέες δράσεις απομειζώντας κάποια κονδύλια από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που είναι ανάλογα με το καθάριστο εθνικό προϊόν. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, κυρίως ε, για μας, γιατί η ουσιαστική πολιτική συζήτηση και οι πραγματικές αποφάσεις για την ε, δημιουργία αυτών των προϋπολογισμών και τη χρήση των κονδυλίων εκφεύγουν του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, εθνικών κοινοβουλίων επίσης. Εκφεύγουν λοιπόν του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Βέβαια εξαρτάται από τη χώρα, γιατί υπάρχουν και διαφορετικές εμπειρίες. Πάντως είναι σαφές ότι οι Υπουργοί Οικονομικών δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξηγήσουν στα κοινοβούλια τους ότι ελήφθη μια χή απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή σε άλλη διεθνή ε, σε άλλο διεθνές φόρουμ, όπως την COP21 για παράδειγμα, για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη π.χ. Και δεδομένου του ΑΕΠ η συνεισφορά μας είναι αυτή. Οπότε πολιτικά είμαστε υποχρεωμένοι να υπερψηφίσουμε αυτή τη συνεισφορά. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Γιατί έχουμε ένα είδος ε, σκιώδους χρηματοδότης, χρηματοδότηση φάντασμα που εκφεύγει οποιοδήποτε κοινοβουλευτικού δημοκρατικού ελέγχου, κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητο. Τρίτον, πρόκειται για ένα θέμα που δεν είχε απασχολήσει μέχρι στιγμής κανέναν. Ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε τα κράτη-μέλη. Ίσως εδώ με διαψεύσουν κάποιοι βουλευτές, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δηλαδή με την εφαρμογή στον προϋπολογισμό της αρχής της επικουρικότητας, γιατί μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής αυτή η αρχή και μάλιστα η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει την δυνατότητα στα Εθνικά Κοινοβούλια να ελέγξουν την εφαρμογή της αρχής αυτής, βγάζοντας κίτρινη ή πορτοκαλί κάρτα, κάτι που έκαναν κάποια Εθνικά Κοινοβούλια πρόσφατα για σημαντικά θέματα. Βέβαια, όταν αποφασίζουμε σε κοινοτικό πλαίσιο, πολύ συχνά και με τη συμφωνία, την έμεση τουλάχιστον συμφωνία των Εθνικών Κοινοβουλίων, με την συμφωνία δηλαδή των κυβερνήσεών τους, που στηρίζονται από κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όταν λοιπόν αποφασίζουμε ότι θα επιφορτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερες ευθύνες σε τομεί κοινών ευθυνών. Δηλαδή θα αυξήσουμε τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Και επίση θα πρέπει να ιδρύσουμε στον τομέα αυτό είτε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, είτε μια διοικητική υπηρεσία, όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κανένας όταν γίνεται μια τέτοια πρόταση, δεν σκέφτεται ότι θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφερθούν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταπεξέλθει στις νέες της υποχρεώσεις. Και γι' αυτό κολλάμε σε ένα αδιέξοδο. Γιατί η απόφαση επί της αρχής που με εντυπωσιακό τρόπο και διατυπατισμούς αναγγέλλεται στο Συμβούλιο, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα μέσα. Είτε είναι ανεπαρκή είτε έρχονται πολύ αργά. Αλλά ακόμη και όταν υπάρχουν τα μέσα, η κατάσταση που δημιουργείται είναι εξή. Εκεί η η θεσπίση συμπληρωματικών κονδύλων είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε οργανισμούς, είτε σε άλλους, άλλες υπηρεσίες, προσθέτει ένα διοικητικό επίπεδο και έσοδα στην, ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό που αυξάνουν όμως και τη φορολογική επιβάρηση των Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε ο φορολογούμενος πάντα πληρώνει σε όλα τα επίπεδα. Τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ήρθε λοιπόν η στιγμή κατά τη γνώμη μας την αρχή της επικουρικότητας στο περιβαλλοντικό να την επεκτείνουμε και στον, στον ε, δημοσιονομικό τομέα. Και έτσι η Ευρώπη με σταθερό ε, δημοσιονομικό κόστος ε, να μπορεί να δρά και όταν ε, ξοδεύουμε ένα ευρώ παραπάνω στις Βρυξέλλες να μην προστίθεται αυτό στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Αντίθετα, να κάνουμε οικονομίες τουλάχιστον ενός ευρώ σε εθνικό επίπεδο. Και μάλιστα, αν γίνεται, να εξοικονομήσουμε πάνω από ένα ευρώ σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, αυτό να σημαίνει η αρχή τη επικουρικότητα. Σε ορισμένου τομεί, η δράση που αναλαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιτρέπει για το ίδιο κόστο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και μάλιστα, να επιτρέπει μερικέ φορέ και σε μείωση του κόστου ή να επιτρέπει αύξηση της αποτελεσματικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η κοινωτική αρμοδιότητα, αλλά είναι και καινή ώρα και είναι σαφές ότι σε θέματα άμυνας, για παράδειγμα, θα έχουμε τη δυνατότητα, δεδομένης και της πολιτικής βούλης που θα πρέπει να διαμορφωθεί, να βελτιώσουμε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολύ μικρότερο κόστος. Σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους στρατιώτες ε, από, από ό,τι οι Ηνωμένε Πολιτείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχουμε 28 διαφορετικού στρατού και μόνο κανένα δεν μπορεί να δράσει. Και όπω έχουμε και Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Εδώ έχουμε δύο τρόπου σκέψη. Είτε να πούμε ότι αυτό που προτίθεται θα προσθεθεί στις εθνικές συνοριοφυλακές και εθνικές ακτοφυλακές, κάτι που είναι παράλογο, ή να πούμε ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε πια ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν ουσιαστικό έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τμήμα ή και το σύνολο των εθνικών τελωνιακών ε, υπηρεσιών ή των εθνικών συνοριοφυλακών και των εθνικών ακτοφυλακών θα πρέπει να αποσπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ίσως δημιουργεί προβλήματα, αλλά αν δεν αρχίσουμε από τώρα να εξετάζουμε και αυτό το πρίσμα του ευρωπαϊκού δηλαδή δημόσιου αγαθού, θα ακινητοποιηθούμε πλήρως, θα παραλύσουμε. Γιατί οποιαδήποτε δράση που η αρχή της θα αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα χρηματοδοτείται και άρα θα καταλήγει σε ανεπαρκείς προσπάθειες ή ε, καθυστερημένες που δεν θα γίνονται αποδεκτές στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, γιατί θα, επιβάλλουν τη θα επιτείνουν τη φορολογική επιβάρηση και τη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα, για παράδειγμα κινητοποιώντα στο δίκτυο των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων ή του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου που θα εξασφαλίζει πλήρη εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και σε δημοσιονομικό επίπεδο και θα επιτρέπει με χαμηλότερο κόστος για το φορολογούμενο, μια αυξημένη αποτελεσματικότητα, γιατί αυτό περιμένουμε όλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαμασούρ. Και εγώ ως πρόεδρος Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, εξετάσαμε ένα σχέδιο αγοράς για ένα κτίριο στο Τόκιο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επίσης ένα μια άλλη πρόταση αγοράς κτηρίου στο Πεκίνο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εκεί δηλαδή που ήδη υπάρχουν 28 πρεσβείες, γιατί κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την πρεσβεία της και στο Τόκιο και στο Πεκίνο. Θα έχουμε όμως επιπλέον μια νέα, 29η πρεσβεία. Έχει νόημα αυτό, δηλαδή θα μπορούσαμε με βάση την αρχή της επικουρικότητας να κάνουμε κοινή διαχείριση ε, των ε, ε, αντιπροσωπιών μας, των προξενείων μας, ή των πρεσβειών μας για τη χορήγηση θεωρήσεων. Οπότε έτσι μπορούμε να αποδείξουμε ότι θα έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ταυτόχρονα θα κάνουμε και οικονομίες. Έτσι θα μπει επιτέλους στο δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει μια πραγματική παγκόσμια δύναμη, μεγάλη δύναμη. Τώρα περνάμε στην άποψη των ακαδημαϊκών. Ε, η κυρία Κωνσταντ Αντόλφ από την Budgets Europe. Πού είναι η κυρία Κωνσταντ Αντόλφ? Έχετε το λόγο για ένα δεκάλεπτο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι κοντά σας ε, και σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί. Με μεγάλη μου χαρά να σας ε, παρουσιάσω δύο μελέτες ε, της Green Budget ε, Europe που είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων. Κάναμε αυτές τις μελέτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι ε, θέμα μας είναι ε, οι είδη πόροι, πράσινοι ήδη και ε, σας είπα, οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν πέρυσι. Ακούσαμε νομίζω σήμερα για δύο θέματα που εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασαν, δηλαδή ο προϋπολογισμός πρέπει να αλλάξει, ο τρέχον προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και το θέμα είναι πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την ε, μετατρεπτική δομή και δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς σας δίνουμε ένα παράδειγμα αυτό που αποκαλούμε πράσινη ήδη πόρη. Εμείς είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι τώρα έχει έρθει η στιγμή των πράσινων ιδίων πόρων. Και θα θέλαμε ε, να σας εξηγήσουμε γιατί πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Αυτό που κάναμε είναι δύο μελέτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις μελέτες αυτές μπορείτε να τις κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας και υπάρχει και κάτι το οποίο κάναμε ε, για το Συμβούλιο Κοφίν της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή ζητήσαμε από τους εμπειρογνώμονες μας να υπογράψουν μια δήλωση ε, και πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη μας χαρά μέσα σε τρεις μόνο ημέρες ε, συγκεντρώσαμε 63 υπογραφές από πολύ σημαντικούς πολιτικούς, πρώην υπουργού οικονομικών, πρώην επιτρόπους και γνωστούς επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα τα πράσινων ιδίων πόρων. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Γιατί τώρα πιστεύουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για τους πράσινους ίδιους πόρους. Μα μιλήσαμε ήδη για το έλλειμμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού και ένα πράγμα το οποίο με εντυπωσιάζει είναι ότι ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που δεν έχει είναι το να καθοδηγεί να δίνει αυτό τον τόνο. Και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την κλιματική αλλαγή. Θέλω να σας εξηγήσω ότι εδώ πρόκειται ε, και για μια κοινωνική και οικονομική ατζέντα και όχι μόνο πράσινη ατζέντα. Τώρα, πράσινοι διπόροι είναι εκείνοι οι οποίοι ε, προσπαθούν, όπως είπα, να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα τροποποίησης του ε, νοσιακού προϋπολογισμού τίθεται το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό αναφέρθηκε και προηγουμένως. Εξετάζουμε την αρχή «Οριπένων πληρώνει». Γιατί στα κράτη-μέλη πρέπει να εκταμιεύονται κονδύλια από το εθνικό προπολογισμό για κάτι που δεν προκαλέσανε τα ίδια τα κράτη-μέλη, αλλά κάποιοι τρίτοι. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για να μην αναφερθούμε και σε καλύτερη ε, εκταμίευση των κονδυλίων. Όπως ε, γνωρίζετε, η παράγραφος 2 της Συμφωνίας ε, του, των Παρισίου μας φέρει, φέρνει στον στόχο του 1,5. Κάτι που ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο του 1,5 γιατί οι πολιτικές μας μέχρι το 2025 και το 2030 εξετάζουν μόνο το 2%. Το πρόβλημα το που δείτε εδώ είναι η UNEP έχει κάνει κάποιους υπολογισμούς και εάν ο κόσμος στο σύνολό του θέλει να πετύχει το 1,5% ε, θα πρέπει οι πολιτικές μας και τα σχετικά κονδύλια να αυξηθούν κατά 20%. Ε, νομίζω ότι αν δεν χρησιμοποιηθούν ε, χρηματοδοτικά εργαλεία όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι δεν πρόκειται για μια προσέγγιση μιας οικονομίας στο σύνολό της, δηλαδή Αυτά αν θέλετε μπορείτε να τα συζητήσετε και τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δηλαδή ε, κατά πόσον οι στόχοι της ε, αηφόρου ανάπτυξης ε, θα αντικατασταθούν μετά το 2020. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί και νομίζω εδώ μπορούν αν διευκρινιστούν αυτά να κερδίσουν όλοι. Τώρα γιατί μιλάμε για πράσινους ήδη πόρους και γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό για τους πόρους αυτούς. Σας είπα υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες ε, που δεν ε, τιμολογούνται στο τι πληρώνουμε εμείς. Ε, εμείς τις τιμές που καταβάλουμε υπάρχουν, καταβάλλονται ενισχύσεις, σημαντικές ενισχύσεις και αυτό θα εξεταστεί στον επόμενο προπολογισμό και σε σχέση με τις εκπτώσεις και σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του προπολογισμού. Κατά τα άλλα θα πρέπει να δούμε λιγάκι αυτά που μας προκαλούν τρίτη κάτι το οποίο είναι πολύ δαπανηρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όσον αφορά το θέμα των ενισχύσεων ε, θα εξακολουθήσει να υπάρχει αυτό γιατί προφανώς και η μετανάστευση δεν σταματάει στα εθνικά σύνορα. Υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια αγατά που έχουν κάποιο κόστος και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αρχίσουμε να το εξετάζουμε. Και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλές δράσεις ε, οι οποίε στο μέλλον θα είναι ιδιαίτερα δαπανήρες Ας δούμε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Αν δούμε λιγάκι τα έσοδα από φόρους στα ε, κράτη-μέλη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι υπάρχει ο φόρος επί του ο φόρος ΦΠΑ, αλλά αυτά βέβαια δεν τα βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια. Αν δούμε λιγάκι ε, τους περιβαλλοντικούς φόρους ε, σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι κάτω από 2%. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει τεράστιο περιθώριο να εξετάσει κανείς ε, και τους δημόσιους πόρους κάτω από αυτό το πρίσμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να επιτευχθούν. Η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν θα αναφερθώ στις επιπτώσεις ε, στην απασχόληση. Αυτό που διαπιστώσαμε στη χρηματοπιστωτική κρίση είναι ότι μόνο οι πράσινοι ε, τομείς μπορούσαν να προσφέρουν ποιοτικές νέες θέσεις απασχόλησης. Έχουμε υψηλό ποσοστό αναργίας ε, και μεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγουμε περισσότερα από 500 δις ευρώ. Ε, αυτό ε, μπορείτε να το συγκρίνετε με τον προεπλογισμό 145 δις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μιλάμε για τρεις φορές επάνω το ποσό αυτό. Ε, και μιλάω, όπως σας είπα, για εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι συνεπάγονται ένα τεράστιο κόστος. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει 10,1% αύξηση στην αναλογία ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς φόρους και φόρους στην εργασία. Αυτό που κάναμε στην πρώτη μας μελέτη είναι ότι εξετάσαμε τέσσερα διαφορετικά εργαλεία, τέσσερις διαφορετικούς φόρους, μεταξύ αυτών και τον ενεργειακό φόρο και εξετάσαμε την περιβαλλοντική απόδοση, κυρίως όμως την οικονομική απόδοση και την κοινωνική απόδοση, όπως επίσης και το θέμα των ενισχύσεων. Και διαπιστώνεται ότι όλα αυτά έχουν ένα ε, τεράστιο δυναμικό για να συμβάλλουν στον ενωσιακό προπολογισμό. Κάποιοι από του φόρους αυτούς μπορούν να συμβάλλουν καλύτερα στον κοινωνικό τομέα, άλλοι στο οικονομικό. Υπάρχουν ακόμα πολλά που υπολείπονται. Ε, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά τα γνωρίζουμε, γνωρίζουμε τους αριθμούς, όμως ε, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουν για όλα αυτά οι εκλογείς και να μιλήσετε και εσείς στο εκλογικό σας σώμα. Έτσι λοιπόν, εξετάσαμε εμείς οκτώ διαφορετικά θέματα και άκουσα ότι ο φόρος ε, στον άνθρακα ε, προτείνεται στην εκθεσιμόντη και το λέμε και εμείς ότι θα πρέπει αυτός να το εξετάσει στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που κάναμε επίση στη μελέτη είναι ότι ορίσαμε διάφορες ομάδες στόχο και μετά εξετάσαμε το πώς μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να απομυθοποιήσουμε όλα αυτά που γνωρίζουμε για την ε, περιβαλλοντική φορολόγηση και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορες ομάδες ε, στόχο. Προφανώς εξετάσαμε οικονομικής φύσεως θέματα, θέματα αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας, ε, κοινωνικά θέματα, θέματα που ενέχουν την κοινωνική αλλά και την περιβαλλοντική διάσταση. Και αυτό που προσπαθήσαμε τελικά να κάνουμε είναι να δούμε ποιο ακριβώς είναι το παιχνίδι της εξουσίας, γιατί είναι τόσο δύσκολο, ε, γιατί ξεκινάμε συνεχώς από θέματα ανταγωνιστικότητας, ενώ γνωρίζουμε ότι κάποια από τα πιο ανταγωνιστικά μέλη ε, όπως η Ινδονία και η Σουηδία, επιπάλλουν όλους αυτούς τους ε, υψηλούς ε, φόρους. Η Δανία είναι πολύ ανταγωνιστική αλλά και η Σουηδία. Αν δούμε λιγάκι το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εδώ και αρκετό καιρό και αυτό το επαναλαμβάνουν συνεχώς οι επιστήμονες, γνωρίζουμε ότι σε σχέση με άλλους φόρους. Ο φόρος επί του εισοδήματος ε, δεν μπορεί να συγκριθεί με το φόρο για το περιβάλλον και νομίζω ότι μόνο αν συνεργαστούμε όλοι, μόνο, θα μόνο τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα θέματα της ε, προστασίας του κλίματος. Για τις ενισχύσεις, τα ακούσαμε αυτά, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη μετανάστευση ε, σε εθνικά σύνορα. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το πλεονέκτημα σε αναδυόμενες οικονομίες. Θα πρέπει και εμείς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλά να σας δείξω τις τελευταίες μου διαφάνειες για το φόρο επί του άνθρακα. Βλέπετε, τα εξετάσαμε τις διάφορες ομάδες αριστερά και προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε κάποια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα για αυτούς τους φόρους επί του άνθρακα. Και εξετάσαμε το ερώτημα το γιατί βλέπουμε να υπάρχουν τόσα πολλά θέματα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις ε, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει σε οικονομίες ε, περιορισμένης χρήσης άνθρακα και χαμηλών ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό έχει γίνει κατά το παρελθόν, θα πρέπει όμως κάπως να επιταχυνθεί. Ή τα θέματα της ε, ισότητας. Ε, όχι. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια θέματα αντιστάθμισης κατά την εφαρμογή αυτών των φόρων. Χωρίς τα εθνικά κοινοβούλια, χωρίς εσάς, χωρίς τους ε, πολίτες, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά αυτά ε, αφορούν την Ευρώπη, είναι γεννή στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, προφανώς και είσαστε κι εσείς ε, στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα κράτη-μέλη που υπέγραψαν τη Συμφωνία Παρισίων ε, και αυτό έχοντας πάντα κατά νου τα θέματα της ανταγωνιστικότητας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πες μου τι φορολογείς και τι δεν φορολογείς και τι δαπανάς και τι δεν δαπανάς και εγώ θα σου πω ποιοι είναι οι πραγματικοί σου στόχοι. Και εύχομαι μετά από 7 χρόνια να μην χρειάζεται πια να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκφράζουν τις προτεραιότητες που σας εξέφρασα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ε, πολύ σαφή παρουσίασή σας, που δείχνει ξεκάθαρα ότι η φορολογική εξουσία είναι στα χέρια των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αν συνέβησαν κάποια σκάνδαλα τύπου LuxLeaks, Panama Papers, συνέβησαν γιατί. Γιατί. Και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Και διασπαθίζουν ένα τμήμα των πόρων τους Και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτόν τον προβληματισμό τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λόγια που είπατε, κυρία μου, που μας αναγκάζουν να προβληματιστούμε πάνω στους στόχους μας, πάνω στο είδος της κοινωνίας που θέλουμε να προωθήσουμε. Και τώρα ε, η κυρία Ντανούζ Νερούντοβα από την Τεχική Δημοκρατία, πανεπιστημιακός. Δέκα λεφτά, κυρία μου. Καλό θα ήταν να περιοριστείτε στα δέκα λεφτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την ε, ε βιωσιμότητα των ε, ευρωπαϊκών οικονομικών. Ε, αυτό το έγγραφο το παρουσιάσαμε το Σεπτέμβριο του 2006 στην ομάδα υψηλού επίπεδου και θα ήθελα να σας πω και τις απόψεις μου, αλλά να κάνω και κάποιους παραλληλισμούς ανάμεσα στι δικέ μα προτάσει και στην έκθεση Μόντι. Η έρευνά μα, ή μάλλον οι προτάσει μα για, την, για μια βιώσιμη χρηματοδότηση για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίζεται, βασίζεται σε δύο λογικέ. Ότι το τρέχον σύστημα των ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεισφέρει στους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, τέθησαν στην Στρατηγική Ευρώπη 2020, για μια ε, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η δεύτερη λογική είναι υπάρχουν κάποια κενά ε, βιωσιμότητας και ήδη οι πόροι υπό τη μορφή ε, ευρωπαϊκής ε, φορολογίας θα μπορούσε να συνεισφέρει στο να μειωθούν αυτά τα χάσματα στη, βιωσιμο, στη βιωσιμότητα. Και αισθανόμαστε τιμή και χαρά που αυτές οι δύο λογικές απεικονίζονται στην έκθεσή μας. Στην έκθεση λοιπόν Θέλουμε κάποια κριτήρια που θα προωθούν την ε, βιωσιμότητα και να καταλάβουμε ε, τους ιδίους πόρους που θα βασίζονται στους ε, φόρους ως εργαλεία για να κλείσουμε αυτό το χάσμα ε, βιωσιμότητας. Πώς το ορίζουμε αυτό το χάσμα. Καταρχάς, έχουμε ε, υψηλότατους φόρους και όλο και αυξανόμενους επί της εργασίας. 53% περίπου τη συνολική φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από το φόρο εισοδήματο. Ε, Εργασία δηλαδή. Δεύτερον, η όλο και μειούμενη σημασία των διορθωτικών φόρων. Ξεκινήσαμε με την περιβαλλοντική φορολογία από 7,2% και τώρα φτάσαμε στο 6,6% και η κατάσταση είναι η ίδια και στον τομέα ε, των καταναλωτικών φόρων. Τρίτο κενό χάσμα είναι ισχυρότερο φορολογικό ανταγωνισμό, λοιπόν, ε, σημαίνει διάβρωση τη φορολογική βάση, ε, μεταφορά των κερδών και τα συνεπακόλουθα σκάνδαλα. Η τέ, το τέταρτο χάσμα είναι η φορολογική συμμόρφωση και οι φορολογικέ απάτε. Μιλάμε για το χάσμα στη συμμόρφωση στο ΦΠΑ, στον εταιρικό φόρο και πέμπτο, το πέμπτο χάσμα είναι ε, μειούμε, προοδευτικά μειούμενα φορολογικά συστήματα. Δηλαδή ένα διαμετική ε, δύναμη του φορολογικού συστήματος όλο και μειώνεται και η κοινωνική ένταξη όλο και αποδυναμώνεται. Εξού και η αυξανόμενη ανισότητα. Επομένως, προτείνουμε στο έγγραφό μας, πέρα από όλα τα ισχύοντα κριτήρια, να βάλουμε και την βιωσιμότητα, το κριτήριο της βιωσιμότητας. Χαιρόμαστε που η απόψη μας για μια αξιολόγηση που να βασίζεται στη βιωσιμότητα απεικονίζεται στην έκθεση Μόντι και ότι η έννοια του τέταρτου πυλώνα, των τεσσάρων πυλώνων μάλλον βιωσιμότητας όπως προτείναμε εμείς, υπάρχει στην έκθεση Μόντι. Μιλάμε για οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική ε, βιωσιμότητα, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και θεσμική ε, βιωσιμότητα. Και η τελευταία η θεσμική βιωσιμότητα τονίζουμε ότι είναι πάρα πολύ ε, αναγκαία. Γιατί χωρί ένα ε, σωστά λειτουργούν ε, νομικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να συλλέξουμε επαρκή πόρους, ε, από φόρου, δηλαδή. Και επομένω, η θεσμική βιωσιμότητα είναι η πιο σημαντική. Σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα. Η οικονομική ανάπτυξη μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο χάρη σε αυτή. Δεν μιλάμε για την ποσοτική ανάπτυξη, αλλά την ποιοτική ανάπτυξη, που είναι η έξυπνη φυσικά ανάπτυξη. Μιλάμε για την δημοσιονομική ε, βιωσιμότητα, για ε, φο, ε, κρατικούς κυβερνητικούς φόρους που να μην είναι επαχθείς, για οικονομική ε, ευημερία. Στην κοινωνική βιωσιμότητα μιλάμε για τη ε, κοινωνική ένταξη, συνοχή, κινητικότητα, για την ευημερία και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρει η στρατηγική του 2020. Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ήδη πόροι τη Ευρωπαϊκής Ένωση, με βάση τους ε, ευρωπαϊκούς φόρους θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη μείωση της μόλυνσης, να προωθήσουν την πράσινη καινοτομία ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στον τομέα της ε, θεσμικής ε, βιωσιμότητα, για το, δεν μιλάω μόνο για τα, ή, τους ίδιους τους φορείς, δηλαδή τα θεσμικά όργανα, αλλά μιλάω για μια δέσμη κανόνων που είναι προϋπόθεση για να υπάρξει αυτή η βιωσιμότητα. Μιλάμε για μια οριζόντια φορολογική εναρμόνιση, για να σταματήσουμε αυτήν την κούρσα προς τα κάτω. Ε, μιλάμε για μια παρεμβολή στους φόρους ή για την δίκαιη κατανομή του, του οικονομικού άχθους μεταξύ των κρατών μελών. Επομένως, γιατί κάποιοι φόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ήδη υπόλοιπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δεν μπορούμε να του χειριστούμε σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε τεράστια κινητικότητα των φορολογουμένων, ε, διάβρωση της φορολογικής βάσης ε, και μεταφορά των κερδών, πρώτο θέμα. Δεύτερο, ε, υπάρχουν εξωτερικά στοιχεία διασυνοριακά που δεν είναι δυνατόν να τα χειριστούμε σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, φυσικά, το να φορολογήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε έτσι τους αντάτες που κάνουν ό,τι θέλουν και πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Και επίσης θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την, τον υπολογισμό της καθαρής θέσης των κρατών μέλων. Γιατί μερικές φορές οι φόροι είναι πολύ δύσκολο να τους ιχνηλατήσουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την καθαρή θέση του κάθε κράτου μέλους. Φορολογική δηλαδή καθαρή Τώρα, πάμε στην έκθεση πιο κάτω και τι βλέπουμε. Το πιο κοινοτόμο σημείο που αναφέρει η έκθεση είναι διαφορετικές, διάφορες επιλογές που έχουμε για τη φορολογική βάση. Τις αναλύσαμε αυτές και θα πρέπει να είναι ένα ε, καλάθι. Και δεν θα πρέπει να είναι ένας και μόνο φόρος, ας πούμε, που θα βασίζεται στους ίδιους πόρους. Εμείς ε, αυτά επιλέξαμε, αυτούς μάλλον ε, τους φόρους ε, αξιολογήσαμε, για να μειωθεί αυτό το, το χάσμα βιωσιμότητας ένα τριπλό CCTV δηλαδή, ε, επίσης ε, φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ε, φόρος άνθρακα και φόρος στο αεροπορικό εισιτήριο με βάση τον άνθρακα. Ε, το CCTV, η διάβρωση της φορολογικής βάσης και μετα... η κοινή ενωπημένη βάση και φορολογία των επιχειρήσεων. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να έχουμε να κλείσουμε το χάσμα, να περιορίσουμε την διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών και θα μπορούσαμε να μειώσουμε το βάρος στην εργασία των φόρων, έτσι. Ε, θα, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε το περιθώριο να μειώσουμε το, τη φορολογία της εργασίας, να λύσουμε το θέμα της ε, φορολογικής συμμόρφωσης και το πρόβλημα της φορολογικής απάτες, κυρίως τη φορολογική, φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Επίσης, εξετάσαμε το πιθαν, την πιθανότητα να μας αποφέρει έσοδα το CCCTB ε, και το κατά πόσο θα μπορούσαμε έτσι να αντικαταστήσουμε εντελώς τον φόρο που βασίζεται στο ΦΠΑ στο, στο ΑΕΠ, στους ίδιους πόρους δηλαδή. Βλέπετε τα αποτελέσματα ότι θα μπορούσαμε με το CCTV να αντικαταστήσουμε πλήρως ε, τους φόρους για όλες τις χώρες με εξαίρεση την ε, Κύπρο. Ενώ αν έχουμε το CCTB, όχι διπλό CC δηλαδή, πάλι θα μπορούσαμε σε πολλά, στις περισσότερες χώρες να έχουμε αρκετούς φόρους, εξαρτάται από την Κύπρο. Ε, με το ΑΕΠ θα μπορούσαμε να κάνουμε μερική αντικατάστασή τους, γιατί ε, μόνο ε, κάποια, 7 δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν πλήρως αυτόν τον ε, φόρο ΑΕΠ. Τώρα, η εισαγωγή αυτή θα μπορούσε να περιορίσει το φορολογικό ανταγωνισμό και να αυξήσει το ρόλο της διορθωτικής φορολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε επίσης να μας βοηθήσει στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και φοροαπηφυγής. Τώρα, το, τη δυνατότητα ε, συλλογής εσόδων μέσω του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, θα μπορούσε να αντικαταστήσει πλήρως τον, το ΦΠΑ για 8 κράτη-μέλη στην πρώτη παραλλαγή ε, και στην δεύτερη παραλλαγή για 12 κράτη-μέλη και σε σχέση με το ΑΕ θα μπορούσε να αντικαταστήσει πλήρως το ΑΕ ε, στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην περίπτωση των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 28 θα μπορούσε να το να αντικαταστήσει για τα 5 από τα 28 κράτη-μέλη. Τώρα, το φόρο του άνθρακα στα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ένταση των εκπομπών άνθρακα αυτή τη στιγμή στο εισιτήριο που πληρώνεις, ας πούμε. Και τα μισά ε, κράτη-μέλη εφαρμόζουν τέτοιο φόρο, ε, άνθρακα στο ευρωπαϊκό εισιτήριο και τα υπόλοιπα όχι. Δεν εξαρτάται όμως από τον, από το όγκο των εκπομπών ο φόρος αυτός. Κάνουμε του υπολογισμού για τη δυνατότητα συλλογή εσόδων έχουμε και ο φόρος αυτός επιβάλλεται ανατόνο εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα, δεν το βλέπετε διάφορα σενάρια και τη δυνατότητα εισπράξεων έχουμε. Και το τελευταίο είναι ο φόρος άνθρακα. Έχουμε εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής ε, τέτοιου φόρου άνθρακα και βλέπετε το δυναμικό τι έσοδα μπορούμε να έχουμε ανάλογα με την τιμή φυσικά που θα επιβάλλουμε ανατόνο εκπομπής διοξίδιου του άνθρακα. Κλείνοντας, και αυτό το τμήμα απεικονίζεται στην έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου. Χαιρόμαστε γι' αυτό παρουσιάζει διάφορες εναλλακτικέ προσεγγίσεις, λύσεις και τρόπους για να εφαρμόσουμε ε, φορολογία με σκοπό για τους ίδιους πόρους και επίσης ε, γίνεται σύνδεση ανάμεσα στα έξοδα και στα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει, μπαίνει και η λογική της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας και των ευρωπαϊκών δημοσίων αγαθών προϋπόθεση για μια μεταρρύθμιση του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει μέσα του εγγενώς το κριτήριο της βιωσιμότητας. Σας ευχαριστούμε κυρία μου για την πολύ μεστή αυτή ανάλυση, τις προτάσεις σας και την εκτίμηση για του τους πιθανούς ιδίους πόρους που μπορούμε να θεσπίσουμε ε, σε σχέση με τις διάφορες πρακτικές των κρατών μέλων. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο σε όσους ε, το ζήτησαν. Σας παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το τρίλεπτο καθένας, το πολύ τρίλεπτο, για να προλάβουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους όσοι το, το ζήτησαν. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Μπρέσκι Γκρέγκορ, συγγνώμη αν δεν προφέρω καλά το όνομά σα. είναι μέλος τη Πολωνικής Γερουσίας και πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, μέλος της ομάδας ε, μεταρρυθμιστών συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Μόντι και την ομάδα υψηλού επίπεδου με τους εμπειρογνώμονές του που εκπώνησαν αυτή την τόσο άρτια έκθεση. Τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής και οι συστάσεις της ε, μας βρίσκουν σύμφωνους σε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, είμαστε υπέρ του ισορροπημένου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική αυτή η ισορροπία ε, στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Επίσης, ε, δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφύγει στις τράπεζες. Άλλο σημαντικό θέμα που χρήζει επισήμανσης είναι η ιδέα και η πρόταση της αναδιάρθρωσης και της απλούστευσης και της αποσαφήνισης ε, του ενωσιακού προϋπολογισμού. Συμφωνούμε λοιπόν και με αυτή την ιδέα. Επίσης ζητούμε ε, την κατάργηση των εξαιρέσεων, των μειώσεων ε, και των επιστροφών για τα έσοδα στην, στο σκέλος των εσόδων. Κάποια βέβαια σημεία της έκθεσης χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες των ε, επιχειρηματιών, των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αναλύσουμε το φόρο που προτείνεται το φόρο άνθρακα υπό το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και οποιαδήποτε παρεμπόδιση περιορισμός αυτής της ανταγωνιστικότητας θα έχει αρνητικές συνέπειες τα υπόλοιπα έσοδα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πολύ διεξοδική ανάλυση αυτής της πρότασης. Εγώ θα προτιμούσα να επικεντρωθούμε στην διερεύνηση νέων πηγών εσόδων και κυρίως στο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι πολύ πιο εύκολη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου και φαίνεται και δικαιότερος. και από τη σκοπιά πολλών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός προς τα έσοδα. Τώρα ως προς τις δαπάνες, τα έξοδα. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τη χρηματοδότηση κάποιων πολιτικών. Και από αυτή την άποψη ο προπολογισμό μας είναι σχετικά άκαμπτος, δεν είναι αρκετά ευέλικτος. Και γι' αυτό είμαι υπέρ της πρότασης της έκθεσης Μόντι να διερευνηθεί η πιθανότητα αναθεώρησης της κοινή γεωργικής πολιτικής και άλλων πολιτικών που απορροφούν α, τις περισσότερες δαπάνες ε, του προϋπολογισμού. Είναι οι πιο δαπανηρές στον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κάρελ Φίντλερ, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Στην ε, Βουλή των Αντιπροσώπων της Τσεχικής Δημοκρατίας, ανεξάρτητος βουλευτής. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όσο άκουγα τις ομιλίες, κρατούσα λεπτομεριακές σημειώσεις και διαπίστωσα κάποιες αντιφάσεις. Ο κύριος Αρτούια, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι το μερίδιο των τελωνιακών δασμών στα κοινοτικά έξοδα μειώνεται. Και γι' αυτό δίνεται, επίσης δίνεται έμφαση στο σεβασμό των περιβαλλοντικών πολιτικών. Και η βιομηχανική μας πολιτική έπρεπε να λάβει υπόψη κάποια περιβαλλοντικά κριτήρια. Το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ είναι ότι έχουμε πολλά αγαθά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζονται στις ευρωπαϊκές αγορές και προέρχονται από χώρες που δεν τηρούν αντίστοιχες αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές με εμά και έτσι έχουν ένα ανταγωνιστικό πλονέκτημα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή της Τσεχίας ε, που παράγει χάλιβα και έχουμε υποστεί τον αθέμητο ανταγωνισμό του κινέζικου χάλιβα που είναι πολύ πιο φθηνός. Η αιμονή μας λοιπόν σε περιβαλλοντικά κριτήρια ναι μεν είναι αξιέπαινη, αλλά θα πρέπει αντίστοιχα περιβαλλοντικά κριτήρια να τηρούνται και από τους εμπορικούς μας εταίρους. Μόνο έτσι να επιτρέπουμε την εισαγωγή των προϊόντων του στην αγορά μας. Αλλιώς θα πρέπει να προστατευτούμε με τη χρήση τελωνιακών δασμών. Γιατί δεν είναι σωστό να λέμε ότι εμείς θα σεβόμαστε τους περιβαλλοντικούς κανόνες ε, και θα το λαμβάνουμε αυτό υπόψη στη βιομηχανική μας παραγωγή. Αλλά χρειαζόμαστε και κάποια προστατευτικά μέτρα απέναντι σε τρίτους που δεν τηρούν αντίστοιχα περιβαλλοντικά μέτρα. Και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει δεόντως την εσωτερική αγορά. Άρα δεν κάνει το καθήκον της, δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή της. Οι τελωνιακοί δασμοί ε, και το ποσοστό τους στη, στον κοινοτικό προϋπολογισμό μας είπατε ότι μειώνεται. Ε, ευκαιρία λοιπόν να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό. Έτσι, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα γίνουν ξαφνικά πιο ανταγωνιστικές. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαστίζεται από ανεργία Επίσης έχουμε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωγής ενώ ταυτόχρονα μας λείπει εξειδικευμένο δυναμικό και έχουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας. Κάτι που δείχνει ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εντάξει. Το παράδειγμα της χαλιβουργίας μας βάζει σε σκέψεις ως προς την εμπορική μας πολιτική. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να να την αναθεωρήσουμε και να αναζητήσουμε κάποια μέτρα προστασίας. Όταν οι Αμερικανοί επιβάλλουν φόρους ή τελωνιακούς δεσμούς πάνω από 250%, εμείς όταν έχουμε 20% μόνο, ε, σκάβουμε το λάκκο μας. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Η Ελισάβετ Τωμά τώρα, Ευρωβουλευτής από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη του εμπειρογνώμων τη Επιτροπής Μόντι που με την πρότασή του μα επιτρέπουν επιτέλου να ε, ξεφύγουμε από το αδιέξοδο ενό συστήματο που είναι αδιαφανέ, γιατί μιλήσαμε για τι μειώσει και επιστροφές, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και ένα ολόκληρο νεφέλωμα χρηματο, χρηματοοικονομικών μέσων και δορυφορικών προπολογισμών, όπω μα το υπενθυμίσατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε. Επίση, ένα άλλο σημείο που οδηγεί στο αδιέξοδο είναι ότι το, το σύστημα αυτό αντιβαίνει πλήρως το πνεύμα των συνθήκων. γιατί οι συνθήκες προβλέπουν οι ίδιοι πόροι να αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων, ενώ οι συνεισφορές των κρατών μελών δεν είναι πραγματικοί ίδιοι πόροι, αλλά πόροι που έχουν ε, συμφωνήσει τα κράτη-μέλη να παρέχουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οπότε έχουμε έναν προϋπολογισμό που κάθε χρόνο αυτοκαταστρέφεται, με χώρες που προσπαθούν να λύσουν ένα γόρδιο δεσμό ε, και έχουν να διαλέξουν μεταξύ της μείωσης των δικών τους κρατικών δαπανών ή της συμφωνίας να μειωθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Δυστυχώ έβγε στο μεταξύ ο Επίτροπο Έτιγκερ, αλλά χαιρετίζω τη βούληση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί υπέρ αύξηση του μεριδίου των ιδίων πόρων στο 50% ευκαιρία του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Χαίρομαι γι' αυτό και επίση χαίρομαι με τον προσανατολισμό ε, τη φορολογία και των δημοσιονομικών θεμάτων ε, σε πιο ε, αξιέπαινου στόχου, όπω είναι η περιβαλλοντική και η στόχη προστασία του κλίματο. Επίση, καλό θα ήταν να κινητοποιήσουμε και επενδύσεις και για κάποιες οικολογικές μεταρρυθμίσεις και στην πολιτική συνοχή. Επίσης, συμφωνώ με τον Τζέχο συνάδελφο που και αυτός έφυγε γιατί αυτό προσπαθούμε να εγκρίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την προσαρμογή στα σύνορα, γιατί δεν έχει νόημα το φόρο του άνθρακα να τον καταβάλουν μόνο οι Ευρωπαίοι και να πληρώνουμε με μείωση της ανταγωνιστικότητά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να επιβάλλουμε φόρους στα σύνορα σε προϊόντα που έχουν υψηλό αποτύπωμα άνθρακα. Επίσης, συμφωνώ με την θέσπιση φόρων τύπου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και επίση να μειώσουμε τους κινδύνου που συνδέονται με την κερδοσκοπία στα χρηματοπιστωτικά. επίσημη είμαι υπέρ τη δίκαιη φορολογία, όπως είπαν οι εμπειρογνώμονε και οι πανεπιστημιακοί. Επίση το πιο σημαντικό είναι το θέμα της φορολογική δικαιοσύνης. Θέλουμε μια φορολογική δικαιοσύνη που βρίσκεται στην καρδιά της συνοχής και του ευρωπαϊκού οράματος, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτό το όραμα. Επίσης, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι πολυεθνικές, αυτές που αποκομίζουν τα περισσότερα κέρδη, είναι αυτές που καταβάλουν και τους χαμηλότερους φόρους και συμμετέχουν πολύ λιγότερο σε αυτή την ε, υποχρέωση τη φορολογική. Να θυμηθούμε το περίφημο 0,005% της, ε, του φόρου που πλήρωνε η Apple στην Ιρλανδία. Κάτι που το επισήμανε και ζήτησε και αντίστοιχο πρόστιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βέβαια, ε, τώρα βρισκόμαστε απλώς στη βάση που δεν λαμβάνει καν υπόψη ε, το σημαντικό πλούτο που δημιουργείται και κυρίως το πλούτο που αφορά το άειλο κεφάλαιο που δεν λαμβάνεται υπόψη στις προτάσεις. Ούτε έχουμε φτάσει ακόμη το ποσοστό που επιζητούμε για τους ίδιους πόρους και ούτε καταφέραμε να εξαλείψουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Και επίσης συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λαμασούρ ότι όταν έχουμε απόφαση για νέα ε, για νέε αρμοδιότητε οι υπάρχουσε πολιτικέ. Ε, εκεί έχουμε μια αποτελεσματικότητα που μπορεί να προκύψει από την επικουρικότητα. Αλλά μερικέ φορέ πρόκειται για νέε πολιτικέ. Για παράδειγμα, για την ενεργεία των νέων, για το σχέδιο οικονομική ανάκαμψη το σχέδιο το επενδυτικό του Γιουνκέρ. Εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα επικουρικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να, βρούμε το κουράγιο και να πούμε κάτι που είναι δύσκολο μερικές φορές, να τολμήσουμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε συστηματικά την μεταφορά κονδυλίων από τον ένα τομέα στον άλλο. Επίσης, σε δημοσιονομικές γραμμέ σημαντικέ, όπω η έρευνα και η καινοτομία, ε, περικόπηκαν κονδύλια και είναι κρίμα να γίνονται τέτοιε περικοπέ. Επίση, τα θέματα της ασφάλειας, ε, όταν βλέπουμε τα ποσά που αφιερώνονται εκεί και όταν γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, αυτές τις μεταφορές από τον ένα τομέα στον άλλο. Εντάξει, έχω και άλλα να πω, αλλά μάλλον θα τα αφήσω για άλλη φορά, μια και με διακόπτετε. Ευχαριστώ κύριε Τωμά. Ο Αλέων Λαμασού θα φύγει σε λίγα λεφτά και θα του δώσω το λόγο, ούτω ώστε να μας κάνει κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες αντιδράσεις μετά από τα όσα άκουσε από του εμπειρογνώμονες και από τους ε, βουλευτές. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, Πρόεδρε. Κάποιες αντιδράσεις και κάποιες απαντήσεις, ενδεχομένως. Μην ξεχνάμε, και είναι κάτι πολύ θετικό, το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας θα μας δώσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να κάνουμε συμπληρωματικές μελέτες, που, κάτι που πρότειναν ορισμένοι, όπως ο πρόεδρος Μπερέσκι, και να συζητήσουμε ο καθένα στη χώρα μα και όλοι μαζί στο Συμβούλιο Υπουργό, Υπουργών Οικονομικών. Γιατί τελικά ποια είναι η ιδέα. Και ποιο είναι ο στόχο, όπω υπενθύμησε και ο Επίτροπο και όπω πρότεινε και η ομάδα υψηλού επίπεδου. Να είμαστε έτοιμοι, ούτω ώστε οι ενδεχόμενε μεταρρυθμίσει επί των οποίων θα συμφωνήσουμε να ξεκινήσουν παράλληλα με το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή από το 2020 και μετά. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη διάκριση ανάμεσα στις, στα νέα έσοδα που θα μπορούσαν να είναι υπέρ του κοινοτικού προϋπολογισμού των 27 κρατών μελών και έσοδα που θα μπορούσαν πιο εύκολα να χρηματοδοτήσουν την ενισχυμένη συνεργασία. Μέχρι στιγμής δημιουργήσαμε λίγες ενισχυμένες συνεργασίες που δεν απαιτούσαν κάποια οικονομικά μέσα. Μεταξύ όμως διαφόρων προγραμμάτων που έχουν ήδη ξεκινήσει ε, είναι κάποιες σημαντικές συνεργασίες, πολύ δάπανες, παράδειγμα χάρη ο φόρος ε, που είπε η κυρία Μπερέση και ο κύριος Στομά ε, επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, εάν προκύψει, εάν τον εφαρμόσουμε, θα χρηματοδοτήσει μάλλον την ενισχυμένη συνεργασία. Παράλληλα, μπορούμε να, να επιβάλλουμε φόρους ε, στα ποσά της ΕΚΤ εάν ε, υπάρχει χρηματοδοτική δυνατότητα της Ευρωζώνης. Αυτή είναι ένα πόρος που θα μπορούσε να πάει ε, στον προπολογισμό. Επίσης, θα πρέπει να διακρίνω ανάμεσα στο τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι άμεσα. Σε μια πρώτη φάση. Σε τρία χρόνια, Φερρυπίν. Και κάτι που το λέω έτσι εντελώ προσωπικά είναι ότι το CCTB, ένα ευρωπαϊκό συμπλήρωμα δηλαδή, ή ένα ευρωπαϊκό κομμάτι δηλαδή, ενός φόρου επί των κερδών και η εναρμόνιση της φορολογικής βάσης, που θα είναι προϋπόθεση, όλα αυτά θα πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε γι' αυτά. Ελπίζουμε ομόφωνα για να εναρμονίσουμε τη φορολογική βάση που δεν είναι εναρμόνιση των ποσοστών, έτσι, των συντελεστών δηλαδή των φορολογικών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε, ούτω ώστε ένα τμήμα να πάει να χρηματοδοτήσει τον κοινοτικό προπολογισμό. Στο μεταξύ θα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται αλλού. Ε, τις συστάσεις του ΩΣΑ και να δούμε και τι γίνεται με τη νέα κυβέρνηση και το νέο κογκρέσο του, τον ΙΠΑ που είναι πολύ ενεργητικό σε αυτό το τομέα. Επίσης, η ε, ηθική εντός αγωγικών φόρη, εγώ έτσι τους λέω. Δηλαδή ο φως του άνθρακα. Έχουν σαν σκοπό να μην φέρουν χρήματα. Να μην φέρουν χρήματα. Όσο υλοποιούν τον ηθικό του στόχο, το να μην μολύνουμε πια, τόσο λιγότερο σημαντικοί θα γίνονται. Έτσι. Πριν μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές μας, θα περάσουν κάποια χρόνια, έτσι. Αλλά αυτό συνέβη και με τους, ε, τελογικούς, με τους τελωνιακούς ε, δασμούς. Στην αρχή χρηματοδοτούσαν διάφορα πράγματα, ας πούμε, αλλά σύν χρόνο σχεδόν εξαφανίστηκαν. Επομένω, όπω είπαν και οι πρόσωποι των ε, γραφείων μελέτη, καλό θα ήταν να έχουμε ένα μπουκέτο προτάσεων, δηλαδή μια πλειάδα προτάσεων και όχι έναν μόνο πόρο. ο πρόεδρο Μπερέσκι πολύ σωστά είπε ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην αναθεώρηση των εσόδων και των δαπανών δεν θα πρέπει φυσικά στις προτάσεις που θα κάνουμε να βάλουμε σε χειρότερη θέση τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τις ξένες εταιρείες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αν ο φόρος του άνθρακα πληρωθεί από, την, από τις εταιρείες που παράγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ζητήσουμε το ισοδύναμο από ξένες εταιρείες ή εταιρείες οι οποίες εισάγουν τα, εξάγουν μάλλον τα αγαθά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εισάγουμε εμεί. Προσοχή σε αυτό που λένε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού αυτή τη στιγμή. Ε, δηλαδή τα αυστηρά, τα καθαρά έσοδα από του τελωνιακού δασμού. Καθαρή τελωνιακή δασμή. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από τη μία στην άλλη να αυξήσουμε του τελωνιακού δασμού. Μπορούμε να αποφασίσουμε να ενισχύσουμε το οπλοστάσιο της ε, εμπορικής μας άμυνας και να βάλουμε, ε, να προωθήσουμε νόμους anti-dumping. Ε, δεν μπορούμε να αυξήσουμε όμως ενή ανοιχτή ε, του τελωνιακού δασμούς. Πριν φύγει ο Αλάν Λαμασού, να, να ρωτήσω το εξή. Αν ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν δημιουργεί κινδύνους με την κατάσταση των συναλλαγών. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο εύκολο να μετεγκατασταθεί από τις ε, χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Έτσι δεν είναι. Πρώτον, αυτό μας λένε οι υπεύθυνοι στον κλάδο. Εγώ δεν το πιστεύω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια θαυμάσια δουλειά επ' αυτού. Τρίτον, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι τα επόμενα χρόνια, κυρίως με τις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε για τον Brexit, το μέλλον του City, οι, οι περίπλοκες σχέσεις που θα δημιουργηθούν σε όλε τι χρηματοπιστωτικέ ροέ, τι επενδύσει, τα προϊόντα, τα χρηματοπιστωτικά μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου, η νέα αμερικανική νομοθεσία που μιλάει για ρύθμιση, απορρίθμιση διαφορών πραγμάτων. Όλα αυτά τα θέματα ε, θα μας οδηγήσουν στο να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα για τον FTT. Φυσικά αυτό αφορά τη δεύτερη γενιά ιδίων πόρων, όχι την πρώτη γενιά ιδίων πόρων, αλλά αυτά τα λέω εντελώς προσωπικά, έτσι προσωπική μου αίσθηση είναι και άποψη. Πολύ ωραία. Ξαναπερνάμε στις παρεμβάσεις των βουλευτών. Αντώνιο Μισιάνη, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και προϋπολογισμού και προϋπολογισμού της Ιταλίας. Ε, εκπροσωπεί το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαμόρφωση του κοινοτικού προϋπολογισμού, του ενωσιακού προϋπολογισμού, ο τρόπος που διαμορφώνεται, ε, οδήγησε στην κρίση. Και επομένω το μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μέλλον του προπολογισμού είναι πολύ σημαντικό για να ανακάμψει το κοινοτικό εγχείρημα. Και γι' αυτό η έκθεση Μόντι είναι μια βάση αφετηρίας, πολύ ενδιαφέρουσα. Και μπορώ να συμφωνήσω. Τα κρίσιμα σημεία του τρέχοντος ε, κοινοτικού προπολογισμού Μα τα υπενθύμησαν. Δεν θα επανέλθω. Θα ήθελα να κάνω κάποιες αξιολογήσεις πάνω στις προτάσεις που για μένα είναι πιο σημαντικές της έκθεσης Μόντι. Φυσικά, συμφωνώ με το στόχο το να αυξήσουμε ουσιαστικά το βάρος των ιδίων πόρων σε σχέση με τις ε, μεταφορές που βασίζονται στο εθνικό εισόδημα, ε, στο ΑΕ και συμφωνώ το να συνδέσουμε τους νέους ιδίους πόρους με τους βασικούς στόχους παρέμβασης των κοινοτικών πολιτικών με ειδική αναφορά ε, την ενιαία αγορά, το φορολογικό συντονισμό και από την άλλη όλη την αλυσίδα ε, Ευρωπαϊκή ε, Ενεργειακή Ένωση, ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, περιβάλλον κτλ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τους πράσινους ίδιους πόρους. Η κατάργηση των μηχανισμών διόρθωσης που είναι εντελώ αδιαφανή και ακατανόητη πρέπει να, οπωσδήποτε να καταργηθούν. Μπήκαν με την πάροδο των χρόνων για κάποια κράτη-μέλη. Ε, επίσης θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή τη επικουρικότητα στην, ε, στο σχεδιασμό του προπολογισμού. Και ένα προπολογισμό ο οποίο θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί με διαφοροποιημένη γεωμετρία, με μεταβλητή γεωμετρία ανάλογα με το πώ διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, η συνένεση των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέοι δείκτε για να αξιολογήσουμε καλύτερα το κόστος και το όφελος, καθώ και το καθαρό όφελος των κοινωνικών πολιτικών. Το καθαρό κέρδο, αν θέλετε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε απλούς αριθμητικού υπολογισμού, έτσι. Τόσα μπαίνουν, τόσα βγαίνουν. Που στρεβλώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες από πολλά κράτη-μέλη καταλαβαίνουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τώρα, κάποιες τελικές σκέψεις. Εάν ο στόχος μας είναι, για τουλάχιστον οι περισσότεροι από μας, αν έχουν στόχο, να ανακάμψει το ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό εγχείρημα, η ιδέα μιας σημαντικής ανάπτυξης του κοινοτικού προϋπολογισμού, που, σήμερα είναι το 1% του ακαθάριστου κοινοτικού προϊόντος, επομένως είναι αμεληταίο, εάν θα πρέπει οπωσδήποτε να ξανασκεφτούμε το θέμα της αύξησης του προπολογισμού. Δεν μπορεί να είναι ταμπού αυτό το πράγμα. Το να έχουμε δημοσιονομική ουδετερότητα και σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, ναι, αλλά δεν μπορούμε να επανεκκινήσουμε την Ένωση αν ο προπολογισμό είναι τόσο περιορισμένος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να επιβαρύνουμε περισσότερο τους πολίτους και τις επιχειρήσεις, γιατί όπως ε, πολύ σωστά είπατε, το να μεταφέρουμε σε κοινοτικό επίπεδο κάποιες πολιτικές μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Υπάρχει και ένα θέμα, το θέμα των ε, εκπομπών και εκεί μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, αν τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εκπομπές για να βρούμε νέους πόρους. Τελευταίο σημείο, και με αυτό κλείνω, η μεγαλύτερη εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων, ούτω ώστε, ή μάλλον ε, η παρέμβαση η οποία γινόταν με τρόπο εντελώς on and off, ε, πότε συμμετείχαμε, πότε δεν συμμετείχαμε. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι, πρέπει οπωσδήποτε να παρεμβαίνουν συνεχώς τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Το λόγο και τώρα ο Νόρμπερ Πράγμαν μέλος του Bundestag, μέλος Επιτροπής Προϋπολογισμών από την Τσεντεού Τσέσου. Κύριε Μπράκμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Äh, Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά σημεία συμπληρώνοντας τα σχόλια των προλαλισσάντων. Είπατε κι εσείς κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία για καλύτερο συντονισμό των εθνικών και των κοινοτικών κονδυλίων, για να αποφύγουμε την διασπάθηση των ε, δημοσίων κονδυλίων. Σίγουρα. Διαρωτόμαστε όμως θα είναι η τελική λύση. Θα πρέπει να μας βοηθήσουν τα εθνικά κοινοβούλια, θέλουμε να επιτύχουμε σε αυτό το διάβημά μας. Επίσης, αν κρατήσουμε τη δομή του CFP, θα πρέπει να ε, κάνουμε έναν επιταετή σχεδιασμό. Να προβλέπουμε δηλαδή τι θα συμβεί την επόμενη επταετία και ποιες θα είναι οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες. κάτι που ίσως μας δημιουργήσει δυσκολίες, γιατί είναι δύσκολο να προβλέψουμε την έκθεση που θα λάβει η μεταναστευτική κρίση ή άλλα θέματα. Και όπως είπατε, τέτοιου είδους δράσεις στο παρελθόν ε, ήταν εκτός ε, συνήθους πλαισίου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο μέλλον θα έχουμε το ίδιο σύστημα. Θα έχουμε βέβαια τέτοιες έκτακτες περιστάσεις, και έκτακτα περιστατικά, αλλά θα χρειαστούμε και ένα έκτακτο σύστημα για να τα αντιμετωπίσουμε. Ή θα αφήσουμε τον επταετή προγραμματισμό και θα υιοθετήσουμε μια βραχύτερη περίοδο προγραμματισμού, μόνο ετή, διετή, ώστε να έχουμε ένα πιο ελαστικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στις απροσδόκητες εξέλιξεις. Επίσης, μιλήσατε για την έμφαση που θα πρέπει να δώσουμε στην ε, ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ας μην ξεχνάμε το κόστος της ε, Ευρωζώνης. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πληθώρα προτάσεων που στόχο έχουν την αύξηση των δαπανών, αλλά δεν είναι έτοιμη να ζητήσει αυστηρή τήρηση των συμφώνων και των διατάξεων που ισχύουν. Μόνο λοιπόν αν υπάρχει η απαραίτητη εμπιστοσύνη, μόνο τότε θα υπάρχουν και πολλές δυνατότητες για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Si, la parole est maintenant à Gérard Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Gérard πρέ. μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Βέλγιο είναι συνεισηγητής για τους ίδιους πόρους. Εν ε, ε, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τα μέλη της ομάδας υψηλού επίπεδου του κύριου Μόντι. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα σχόλιά τους και πολύ άρτια τεχνικός. Δεν θα σας ε, εκπλήξει το γεγονός ότι είμαι υπέρμαχος και μάλιστα ενθουσιώδης ε, του, της αναθεώρησης του συστήματος των ίδιων πόρων, φυσικό άλλωστε γιατί είμαι και εισηγητής για το θέμα αυτό, με όλου τους, τους διορθωτικούς μηχανισμούς, με όλες τις μειώσεις και τις επιστροφές, με τη δημιουργία την ε, αθέμητη, αθέμητων ε, συμπληρωματικών πόρων και με την αρχή της την αντίφαση ως προς την αρχή της συνθήκης επιστροφής μας δημιουργούν ε, έναν μη βιώσιμο προϋπολογισμό. Θέλουμε λοιπόν μια αναδιάρθρωση και ε, έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα μας κάνει ικανούς να ε, υλοποιούμε τους στόχους μας. Όπως υπενθύμησαν ε, και οι προλαλήσαντες. Ε, η δημοσιονομική κυριαρχία δεν είμαστε εμείς, αλλά εσείς. Όταν συζητούμε τους ίδιους πόρους ε, και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τις κυβερνήσεις και κυρώνονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπότε η επί της ουσίας συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τα εθνικά κοινοβούλια για μια πληθώρα τομέων. Ένα από αυτά τα θέματα, ένας από αυτούς τους τομείς, ε, ε, επί τη ευκαιρία της συζήτησης των ιδιών πόρων, ε, που θα επηρεάσει πολύ και την πορεία των συζητήσεων, είναι το εξή. Σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, μερικά κοινοβούλια απάντησαν, αλλά όχι όλα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων ότι στο μέλλον 50% των κοινοτικών κονδυλίων θα προέρχονται από ιδίους πόρους και οι εθνικές συνεισφορές δεν θα ξεπερνούν το 50%. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ως προς αυτό το στόχο. Δεύτερον, πριν από λίγο ο πρόεδρος μας υπενθύμησε το εξής. Ο κανόνας ε, του ανώτατου του ορίου του 1% ε, του κυρωτικού προϋπολογισμού ως προς το ε, είναι ιερός και απαράβατος κανόνας ή επιδέχεται διαπραγμάτευση ή είναι ένας κανόνας το ανώτατο το 1% ιερός απαράβατος και θα πρέπει να παραμείνει ακέραιος και ανέπαφος. Τρίτον, όπως είπαν και οι εμπειρογνώμονες, το νέο σύστημα ιδίων πόρων δεν μπορεί να δράζεται σε ένα και μόνο πόρο. Θέλουμε ένα καλάθι πόρων. Γιατί χρειάζεται ένα καλάθι πόρων για τουλάχιστον τρει-τέσσερις λόγους. Καταρχήν, οι πόροι δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Το έχουν αποδείξει αυτό οι εμπειρογνώμονε. Όπως μας υπενθύμησε και ο κύριος Λαμασούρ, έχουμε φόρου που ε, είναι αυτοκαταστροφικοί. Όσο πιο αποτελεσματικοί είναι, τόσο λιγότερα έσοδα αποφέρουν. Τρίτον, υπάρχουν ήδη πόροι που θα πρέπει να έχουν μια θετική εξελικτικότητα, δηλαδή να αυξάνονται προοδευτικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται ε, να προσθέτουμε τακτικά νέους, φόρ, νέους πόρους. Οπότε η σύνθεση του καλαθιού αυτού θα είναι εξαιρετικά σημαντική για τον κυρωτικό προπολογισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει συζήτηση και από αυτό, επί τη ουσία με τα εθνικά κοινοβούλια, για το ποιο θα είναι ο χαρακτήρα, η φύση και η εσωτερική ισορροπία αυτού του καλαθιού των πηγών ιδίων πόρων. Άλλο θέμα. Ο ρυθμός εισαγωγής και ο τρόπος εισαγωγής του νέου συστήματος των ιδίων πόρων. Το είπατε κι εσείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του έτους θα υποβάλει νέες προτάσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα καθορίζει για την επόμενη επταετία το ύψος των επιτρεπόμενων δαπανών. Κάτι που είναι υπερβολικός περιορισμός γιατί έτσι θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε σε έκτακτες ή κατεπίγουσες καταστάσεις. Και θα έχουμε και τον Brexit αν επιβεβαιωθεί. Ποιε θα είναι οι συνέπειε τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκ πρώτη όψεω και με βάση τα στοιχεία που κυκλοφορούν, θα έχουμε μείωση των διαθέσιμων εσόδων περίπου 10 δισεκατομμύρια. Με βάση τα στοιχεία που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Οπότε, πώ θα αντιμετωπίσουμε, θα αντισταθμίσουμε αυτή τη μείωση κατά 10 δισεκατομμύρια, είτε θα μειώσουμε τι δαπάνε, κάτι που δεν προτιμώ εγώ, ή θα ε, ανατροφοδοτήσουμε ε, τον προϋπολογισμό. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα 7 δισεκατομμύρια που θα, δεν χρειάζεται πια να καταβάλουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε δεν είναι 10 δισεκατομμύρια που θα πρέπει να βρούμε. Πάντως αυτά τα 10 δισεκατομμύρια που λείπουν από την αρχή θα πρέπει να ανατροφοδοτηθούν στον προπολογισμό από ένα νέο ιδιοπόρο ή από ένα πακέτο ιδιών πόρων ώστε να μην χρειαστεί να αυξήσουμε τις εθνικές συνεισφορές, τις συνεισφορές από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις χώρες ό,τι αφορά τη δημοσιονομική επιβάρηση και τον δημοσιονομικό προσανατολισμό τους. Επίσης, ε, συμπληρωματικά έσοδα που στο μέλλον ίσως αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Τα εθνικά κοινοβούλια συμφωνούν ότι τα έσοδα που απορρέουν από την εφαρμογή των αμυγός κοινοτικών πολιτικών, για παράδειγμα την πολιτική ανταγωνισμού και το σεβασμό των κανόνων του ανταγωνισμού. Εδώ, μετά από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επιβάλλονται πρόστιμα. Θεωρείται θεμητό τα πρόστιμα αυτά και τα έσοδα που προέρχονται από την εφαρμογή των αμυγός κοινοτικών πολιτικών να ενταχθούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, θα έχουμε ένα νέο σύστημα ε, Προκατακτική ε, άδεια για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Το σύστημα αιτία, όπω το έχουν και οι Αμερικανοί. Οπότε ο κόσμο θα πρέπει να πληρώνει. Γιατί το σύστημα αιτία θα ε, έχει κεντρική διαχείριση. Μπορούμε αυτά τα έσοδα να τα ε, εισαγάγουμε στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και κάθε φορά που έχουμε μια ειδική αμυγός κοινοτική πολιτική Πού δημιουργεί έσοδα. Αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα τροφοδοτούν τον κοινοτικό προπολογισμό ως συμπληρωματικός πόρος. Ίδιος. Αυτά. Γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο και τώρα ο κύριος Σέξιν. Μάλλον ε, κάπως διαφορετικό είναι το όνομα από την Πολωνική Βουλή μέλος του ECR και μέλος Επιτροπής ε, Δημοσιονομικών της Πολωνικής Βουλής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, λέει ο κύριο Σάσιν, για την ευκαιρία που μας ε, δίνετε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση επί της εκθέσεως Μόντι. Θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο Μόντι για το σημαντικό αυτό πόνημα και τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της πολύ σημαντικής και ενδιαφέρουσας έκθεσης. Έχουμε πολλά συμπεράσματα ε, της έκθεσης που μας βρίσκουν σύμφωνους. Για παράδειγμα, η κατάργηση των διορθωτικών μηχανισμών, των rebates, των επιστροφών και μειώσεων. Γιατί ε, έτσι θα ενισχύσουμε τη διαφάνεια του κοινοτικού προϋπολογισμού. Και η κοινωνία ε, των κρατών μελών θέλει να καταλάβει πώς διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός. Γι' αυτό και θέλουμε έναν ευανάγνωστο, εύληπτο και ε, σαφή, διαφανή προπολογισμό. Είναι σημαντικό ο προπολογισμό να είναι διαφανή. Επίση, ε, η αναζήτηση νέων πηγών ιδίων πόρων. Συμφωνούμε με μερικέ προτάσει τη έκθεση Μόντι. Για παράδειγμα, είμαστε υπέρ του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θεωρώ ότι είναι πολύ δίκαιη αυτή η πρόταση και σίγουρα ε, άξια να, διερευνηθεί. Έχουμε κάποιους δισταγμούς για το φόρο του άνθρακα. Όχι ως προς την ανάγκη διαφύλαξης ε, της ε, α, ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος, είναι θέμα κοινοτικής αλληλεγγύης. Ε, η κοινοτική αλληλεγγύη είναι από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχουμε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των χωρών μελών, ε, και εξαιτία τη ιστορική εξέλιξη τη οικονομία τους ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτέ οι διαφορέ. Η πολωνική οικονομία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στον άνθρακα που είναι η βασική πηγή ενέργειας και πολύ φοβούμαι ότι αν ε, πιέσουμε για αυτή τη λύση του φόρου του άνθρακα θα, <laughs> θα, θα προταθεί αναζωογόνηση των διορθωτικών μηχανισμών, των rebate και των επιστροφών, γιατί με τέτοιες διαφορές θα ανακύψει και πάλι η ανάγκη επαναφοράς των διορθωτικών μηχανισμών, αν ε, επιβάλλουμε μέτρα από το φόρο του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε όλες αυτές τις προτάσεις. Επίσης το θέμα του αθέμητο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες ε, που δεν σέβονται τόσο αυστηρές περιβαλλοντικές διατάξεις με εμάς. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προϊόντα αυτών των χωρών. Επίσης, τι συγκεκριμένες διατάξεις ε, μπορούμε να επιβάλλουμε για τα προϊόντα αυτών των χωρών. Για να μην έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Και θα πρέπει επίσης πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε όλο το θέμα των τελωνιακών δασμών και του ύψους τους, όπως πρότεινε και ο κύριος Λαμασούρ. Σας ευχαριστώ. Βέβαια, αλλά ο φόρος άνθρακα στα εξωτερικά σύνορα ίσως ε, θα μπορούσε να αντικαταστήσει σε κάποιο βαθμό ε, τα, τους τελωνιακούς δασμούς. Τώρα, ο κύριος Μάρκα, από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση, σοσιαλιστής μέλος Επιτροπής Οικονομικών και μάλιστα και γενικός συζητητής στη σχετική έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, καλεσμένους ε, που μας διαφώτισαν ε, για τις συστάσεις της έκθεσης Μόντι, τις συστάσεις ε, της ομάδας υψηλού επίπεδου και χαίρομαι για τις προτάσεις που, και τα σχόλια που δείχνουν μια συνένεση και ως προς τη διάγνωση και ως προς το φύλλο πορείας, ως προς τις προσανατολισμούς και τις δηλώσεις βουλήσεως για την διαμόρφωση του κοινοτικού προπολογισμού. Από τη δήλωση βούλησης βέβαια μέχρι την εφαρμογή, την αυτή εφαρμογή έχουμε μακρύ δρόμο και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε και συγκεκριμένες διευκρινήσεις και να προβληματιστούμε για πολλά θέματα. Τώρα, ως προς την ουσία, σίγουρα οι προθέσεις είναι αξιέπαινες γιατί θέλουμε με παρόμοια μέσα να ε, εντείνουμε την αποτελεσματικότητά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να κάνουμε κάποιες οικονομίες σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά μας χαροποιεί αυτή η πρόθεση. Ε, μας λέτε θα έχουμε καλύτερο προσανατολισμό των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς πολιτικές με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Διαρωτόμαστε λοιπόν. Ποιε θα είναι οι μεταφορέ που θα γίνουν ε, στον κοινοτικό προπολογισμό και σε ποια προγράμματα θα γίνουν οι οικονομίες. Αυτό δεν διευκρινίζεται. Επίσης κάποια πιο τεχνικά ζητήματα, γιατί ένα από τα ζητήματα που μας προβληματίζουν είναι η προβλεψιμότητα των εθνικών συνεισφορών στον κοινοτικό προπολογισμό. Στην περίπτωση της Γαλλίας, για παράδειγμα, διαπιστώσαμε ότι το 2013 είχαμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τις προβλέψεις και για άλλες χρονιές είχαμε ένα... 2 ε, δισεκατομμύρια λιγότερο, τεράστιες διαφορές δηλαδή μεταξύ των προβλέψεων και των αναγκών. Το θέμα της προβλεψιμότητας λοιπόν και της διευκόλυνσης ε, της δημοσιονομικής εξέτασης στα κράτη-μέλη λαμβάνεται υπόψη στους ε, στόχους που καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Επίσης υπάρχει και το θέμα της δίκης επιστροφής. Το επισημάνατε, το αναπτύξατε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εξηγήσουμε καλύτερα στους Ευρωπαίους πολίτες τι νομιμοποιεί τη δράση μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπουν σχετικές εργασίες για το 2017 και ποιοι θα ήταν οι βασικοί δείκτες που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί για να εμπλουτίσουμε αυτή την ανάλυση και να έχουμε πιο άρτια επιχειρηματολογία προς την κοινή μας γνώμη για να μπορέσουμε ε, να πείσουμε πιο αποτελεσματικά τους Ευρωπαίους πολίτες για το ενδιαφέρον ε, και την ανάγκη χρηματοδότησης του κοινοτικού προγράμματος. Ε, κύριε Σαμασούρα, έφυγε. Φαντάζομαι ο κύριο Κάρφιν θα απαντήσει. Η ομάδα υψηλού επίπεδου για του ίδιους πόρους, δεν ε, ενέκρινε την πρόταση φόρου ή τέλους για τις οδικές μεταφορές στα πλαίσια της οδηγίας για τις ευρωβινιέτες ή μια για το φόρο στα... στις... στις αεροπορικές μεταφορές, φόρο στα αεροπορικά εισιτήρια. Γιατί αποκλείστηκαν αυτοί οι δύο φόροι στις οδικές μεταφορές και στις αεροπορικές. Η απόρριψη οφείλεται σε τεχνικούς ή σε πολιτικούς λόγους στο κατά πόσο δηλαδή θα γίνουν πολιτικώ αποδεκτά αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Για την προβλεψιμότητα, να σας πω ότι υπάρχει μια στρέβλωση ανάμεσα στις δεσμε... ανάληψη δεσμεύσεων και στις πιστώσεις πληρωμών. Οι συνεισφορές των κρατών μελών βασίζονται στις πληρωμές. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης που ψηφίσουμε κάθε χρόνο ε, ε, βασιζόμαστε στις ε, δεσμεύσεις ανάληψη υποχρεώσεων 157,8 ε, δισεκατομμύρια. Οι πληρωμές είναι 130 δισεκατομμύρια. Οι πληρωμές δεν είναι κάτι που ζητάνε τα κράτη-μέλη. Σαν να υπάρχει καθυστέρηση στην ε, έναρξη των διαφόρων προγραμμάτων. Είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί. Και εδώ ζητάω από τους ε, εθνικούς ε, βουλευτές και μέλη των ε, Επιτροπών Προϋπολογισμού και Οικονομικών να σας ρωτήσω το εξής. Ε, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα κράτη-μέλη γιατί οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις δεν καλύπτουν το 100% των προγραμμάτων. και μερικές φορές βλέπουμε, βλέπουμε μάλλον από χρόνο σε χρόνο πόσο υπαναχωρούν τα κράτη-μέλη από διάφορα προγράμματα γιατί δεν μπορούν να συμπληρώσουν το ποσό που υπολείπεται. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Ε, είναι τόσο περίπλοκοι ε, οι διαγωνισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να απεμπλακούν οι πιστώσει. Άραγε, διερωτώ, διερωτώμεθα, γιατί κάθε χρόνο μα επιστρέφουν χρήματα τα κρατημέρια. Και τα κράτη-μέλη επιστρέφουν κάποια κονδύλια, γιατί αντίθετα από αυτά που είχαμε προβλέψει, δεν ε, υπήρξαν οι απαραίτητε πιστώσει. Δυσκολία είναι αυτό, τεράστιο. Γιατί η Ευρώπη θέλει να ενθαρρύνει τι επενδύσει και κάθε φορά που ξεκινάμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επί δύο ή τρία χρόνια δεν ξεκολλάει αυτό το πράγμα, δεν απογειώνεται. Και έχουμε ένα φαινόμενο γιογιό πάνω κάτω πάνω κάτω, όπως έλεγε ο κύριος Ντεπρέ. Δηλαδή, στην αρχή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου έχουμε λίγες πληρωμές και στο τέλος του πλαισίου, έτσι, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ξαφνικά έχουμε αιτήματα, ας πούμε, ε, και αδυναμία πλήρωση, πληρωμών, όπως συνέβη και στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, το 2013-2014, α πούμε. Το, το λέω αυτό εντός παρενθέσεω. Ο Βλαντιμίρ Μάνκα ε, τώρα ε, που είναι μέλος των σοσιαλιστών, της ομάδας των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν σε πάρα πολλά κράτη εθνικά ελλείμματα και αυτά οδηγούν στο ότι ε, αυξάνεται ο αριθμός ε, των κρατών όπου η Κομισιόν διαπιστώνει ότι υπάρχει καθυστέρηση στις ε, πληρωμές. Ε, το σύστημα ε, το οποίο επιτρέπει κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο όπου υπάρχει αυστηρός ε, προγραμματισμός. Και μετά έρχονται οι δήμαρχοι και λένε ότι υπάρχουν καθυστερείς πληρωμές αλλά μερικές φορές το προκαλούμε μόνοι μας. Αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί καλά και γι' αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από δύο χρόνια πιέσαμε το Συμβούλιο να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για τη Frontex. Ε, τους είχαμε πει ότι το θέμα επήγει και το Συμβούλιο είπε όχι. Και όταν επήλθε η καταστροφή τότε το Συμβούλιο ε, αύξησε ε, κατά τρεις φορές τα κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν το σύστημα δεν είναι καλό και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που η ομάδα Μόντι, όπου συμμετέχει και ο κύριος Κάλφη και ο κύριος ε, Λαμασούρ. Ε, χαίρομαι που αυτή η ομάδα έχει επεξεργαστεί ένα πολύ καλό έγγραφο και χαίρομαι και για αυτά που αναφέρετε εσείς εδώ ως πράσινο προϋπολογισμό εκείνοι οι οποίοι εισάγουν από τρίτες χώρες και όταν ε, προκύπτουν ε, υψηλές εκπομπές, ε, αυτοί φορολογούνται, πρέπει να φορολογούνται και με τον τρόπο αυτό θα παραμείνουν και οι δικοί μας η παραγωγοί ανταγωνιστική. Αλλιώς θα εκδιωχθούν από την αγορά και θα έχουμε και ένα πολύ καλό εργαλείο για την προστασία του κλίματος. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον μας. Οι πολίτες έχουν πραγματικά το αίσθημα ότι τους αφαιρούμε κονδύλια από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. ότι αυτά τα κονδύλια μπαίνουν στον ενωσιακό προπολογισμό. Ε, δεν ξέρουν βέβαια ότι πάρα πολλά χρήματα τους επιστρέφονται μέσα από τις ενισχύσεις που λαμβάνουν. Ο κύριος Λαμασούρ είπε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μία αποτελεσματικότητα στο όλο σύστημα, να υπάρχει μία κοινή, αν θέλετε, πολιτική άμυνας ε, γιατί αν κάνουμε από κοινό αγορές, ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε μέχρι και 100 δι ε, ευρώ, που μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ε, ποσό. Α ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό τον δρόμο. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε έναν ευφυή e, ενωσιακό προπολογισμό, όπου οι άνθρωποι θα έχουν την αίσθηση ότι οποτεδήποτε καταβάλλονται κονδύλια σε αυτό τον κοινό κορβανά, προκύπτει και εξοικονόμηση. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Φτάσαμε στο τέλος των παρεμβάσεων των παρόντων βουλευτών. μα δω, υπάρχει κάποιος άλλος που ζητάει το λόγο. Όχι. Και τώρα, θα ζητήσω πρώτα από τον κύριο Κάλφιν να μας κάνει τις δικές, τους παρατηρήσεις, τις δικές του παρατηρήσεις, αντιδράσεις και απαντήσεις, τα όσα άκουσε, από τους εμπειρογνώμονες καταρχήν, και να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών. Θέλετε το λόγο. Θέλει κάποιο το λόγο. Τι παρέχει. Ο Γιώργεν Άντερσον, μέλος Επιτροπής Οικονομικών του Σουηδικού Κοινοβουλίου. μέλος του Μετριοπαθούς Κόμματος, το οποίο ανήκει στο, στην οικογένεια του ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ. Ίσως ε, θα μπορούσα να πω κάτι για το ότι η Σουηδία έχει λιγάκι διαφορετική προσέγγιση. Δεν θέλω βέβαια να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ε, το θέμα είναι ότι εμείς δεν διαφωνούμε με το ενωσιακό πρόγραμμα. Κάθε άλλο ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί ε, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Επίσης θέλω να σας πω ότι το θέμα μας δεν είναι το, να, το ότι αντιμετωπίζουμε με επιφυλακτικότητα τους ίδιους πόρους. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, και δεν θέλουμε να προβάλλουμε μόνο τα δικά μας τα συμφέροντα. Υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η Σουηδία, παραδείγματο χάρη, έχει το μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή ανά τον κόσμο και οποτεδήποτε λαμβάνονται αποφάσεις εμείς ε, συμμετέχουμε, ξέρετε, έχουμε μια ευημερούς οικονομία παρά τους υψηλούς φορολογικούς ε, συντελεστές. Γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει κανείς να συνυπολογίζει και επ' αυτού ε, έχουμε πολλά καλά παραδείγματα στη Σουηδία. Βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Εγώ ε, θεωρώ και εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Γιατί να, αποδεικνύεται. Η Σουηδία είναι ανοιχτή. Ανοιχτή έναντι του ε, ελεύθερου εμπορίου, περισσότερη κοινή αγορά, καλύτερη κατανομή των περιουσιακών αξιών και παρόλα αυτά τα καταφέρνουμε μια χαρά. Στην βιομηχανία μας βλέπουμε υπάρχει και αλλαγή των υποδομών. Τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να καταλήξω στο ότι μερικές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι ο ενωσιακός προπολογισμός είναι τεραστίου μεγέθους. Ε, ε, αναφέρθηκε όμως και το ποσοστό 1% και αναφέρθηκαν και οι εκπτώσεις ε, που χορηγούνται πάση περιπτώσει, ο ενωσιακός ε, προϋπολογισμός ε, είναι το 1% και δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι με αυτό το 1% ε, μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου μια πληθώρα θεμάτων, το πώς μπορεί να ορθοποδήσει η οικονομία, Βεβαίω η λύση δεν είναι μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Η λύση δεν είναι επίσης να επιβληθούν νέοι φόροι. Αυτό σίγουρα δεν είναι η λύση. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε έτσι ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τη χρησιμότητα ε, του περιορισμού της ε, γραφειοκρατίας. Και πρέπει επίσης ε, να σκεφτούμε να δούμε ποιοι φόροι πρέπει να εφαρμόζονται. Γιατί οι επιπτώσεις σε κάθε χώρα είναι διαφορετικές και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε όσον αφορά παραδείγματο χάρη στο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ο φόρο αυτό έχει επιπτώσει και σε άλλε χώρε και αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε. Η Ευρώπη ε, δεν είναι ομοιόμορφη, οφείλουμε να σεβόμαστε την ετερογένεια και δεν μπορούμε να έχουμε κατά νου μόνο ο καθένας τα δικά του συμφέροντα. Ε, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία αλλά πολλές φορές ε, γίνεται λόγος για αύξηση του φόρου και των φορολογικών συντελεστών και όλοι λένε ότι θέλουν να ελέγχουν καλύτερα τα ενωσιακά κονδύλια. αλλά ξέρετε, κατ' ουσίαν άλλα λένε και άλλα εννοούν. Και αυτό εμφανίζεται πολύ συχνά και νομίζω λέει πολλά. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ε, ακριβώς ε, ε, οφείλουμε να συζητάμε με τους πολίτες, τι στόχους επιδιώκουμε και να σκεφτούμε και ποιο είναι σήμερα το ενωσιακό εγχείρημα, ποιος είναι ο τελικός μας στόχος. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια, διαφάνεια. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο το οποίο κατανοούν και οι πολίτες και το οποίο το στηρίζουμε όλοι μας. Αν αυτά τα οποία λέμε αποκλίνουν ουσιαστικά από αυτά τα οποία πράττουμε, υπάρχει πρόβλημα. Αυτά είχα να σας πω και εγώ και νομίζω ότι υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά Ελπίζω ε, να τα καταφέρουμε από κοινού στο πλαίσιο του ενωσιακού εγχειρήματο, να βρούμε τη σωστή πορεία, να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη και την, ε, τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στο σύνολό του. Βεβαίως οφείλουμε να επιτύχουμε ανάπτυξη και να αυξήσουμε τον ενωσιακό προπολογισμό, ε, καταβάλουμε περισσότερα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος όλων των κρατών. Και οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς μπορούμε να προκαλέσουμε ανάπτυξη και να εισρέψουν στον ενωσιακό προβληματισμό περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κ. Κάλφιν. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Μέσα στο 2016, πριν από λίγους μήνες, μια άλλη ε, διακοινοβουλευτική διάσκεψη συζήτησε αντίστοιχα θέματα με αυτό το ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Έχω μια καλή αίσθηση από τη σημερινή συζήτηση. Με έκπληξη το διαπιστώνω. Υπάρχει περιθώριο για συνένεση. Αλλά ο σημερινός εθνικός προπολογισμός δεν είναι αρεστός ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ξεχνάτε, να εποπτεύουμε για το πού πάνε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η ιδέα λοιπόν της βελτίωσης του προπολογισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, καλύτερα αποτελέσματα, πιο μεγαλύτερη ευελιξία, είναι κάτι που δημιουργεί περιθώριο, χώρο για περαιτέρω συζητήσεις και ενδεχομένως τελικά συνένεση για το πού πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Πρόεδρε, στην έκθεσή μας εξηγούμε γιατί πρέπει να αλλάξει ο προπολογισμό και πώς πρέπει να αλλάξει. Εξηγούμε αυτή τη λογική. Έχουμε βάλει διάφορα πιθανά σενάρια, ε, διάφορες πηγές εσόδων. Κάποιες από αυτές σας παρουσιάστηκαν. Μια θαυμάσια ανάλυση των ακαδημαϊκών και των ειδικών. Ακούσαμε κατ' επανάληψη ότι εμείς στη δική μας ομάδα, ε, στην ομάδα Μόντι, ε, τέτοιες παρουσιάσεις ακούσαμε κατ' επανάληψη και προσπαθήσαμε αυτές τις λογικές να τις ε, ενσωματώσουμε στην έκθεση. Η βασική λογική είναι ότι δεν καθορίζουμε τις πηγές των επιπρόσθετων πόρων, ε, απλώς υποδεικνύουμε κάποιες πιθανές πηγές, πώς μπορούν να συνδυαστούν, ποιο είναι το καλάθι από το οποίο θα προέλθουν τα έσοδα αυτά. Α, όλα αυτά είναι προσυζήτηση. Φυσικά το καλύτερο είναι να δημιουργήσουμε αυτό το, το καλάθι, ούτως ώστε να επηρεάζει με δίκαιο τρόπο τα κράτη-μέλη και να βαραίνει με δίκαιο τρόπο τα κράτη-μέλη και το καλάθι αυτό θα πρέπει να συνδέεται με την αξία που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα καθήκοντα τα οποία προσπαθεί να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση και στις προτάσεις μας. Ο συνδυασμό και οι ειδικέ πηγές από το που θα υπάρχει ας πούμε ε, φόρος ή, που δεν θα υπάρχει ας πούμε, ο δικός φόρος, ερώτηση που έκανε ο κύριος Φρανκ, αυτά είναι θέματα που θα λυθούν στην πορεία. Μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα σενάρια, διάφορες πιθανές πηγές, διάφορους συνδυασμούς. Πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα που ακούστηκαν. Να απαντήσω σε αυτές. Θέλω να υποστηρίξω αυτά που ο κύριος Μιστάνη, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε δείκτες για ε, και να αντικαταστήσουμε το, την προσέγγιση καθαρών εσόδων. Δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε την, ε, την καθαρή θέση μιας χώρας. Δεν είναι καμία χώρα η οποία μπορεί να ποσοτικοποιήσει σε χρήματα, ας πούμε, τα εφαίλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρότι ακούστηκαν κάποια παραδείγματα, ακούστηκαν άλλα παραδείγματα από την Πολωνία, Φερρυπίν, ότι κάθε ευρώ που ε, επενδύεται στις πολωνικές ε, υποδομές, το 50% καρπώνονται οι Γερμανοί από αυτό το ευρώ. Δεν μπορεί να μπει έτσι, με λογιστικούς όρους. Όταν μιλάμε για καθαρή θέση, όταν μιλάμε, ως με το μεγαλύτερο λιμάνι, το θαλάσσιο λιμάνι είναι ε, στο Ρότερνταμ, ε, αυτό συνδέεται με την ε, ύπαρξη της ενιαίας αγοράς, εξού και η σημασία αυτού του λιμανιού. Γι' αυτό παίρνει και, ε, έχει και τέτοιο τζίρο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούν να δοθούν. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε πόσα δίνουμε, πόσα παίρνουμε να πούμε τριστολάδι, τριστοξίδι. Παράλληλα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη, α την πούμε, ή ξέρω, πέστε την δείκτε, ούτω ώστε να επικοινωνήσουμε. Γιατί πραγματικά οι πολίτε πρέπει να ξέρουν ε, τι παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά τι πληρώνουν για να τα πάρουν όλα αυτά. Φυσικά δεν είναι ταμπού για το να μιλήσουμε για το μέγεθο του προπολογισμού, αλλά αυτό δεν είναι το, ο σκοπό τη έκθεση. Επίτηδε αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε για τον όγκο, για το, τα ποσά του, του προπολογισμού. Και γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί στα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξουν αλλαγέ. οπωσδήποτε. Μία από αυτέ θα είναι ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Ή τέλο πάντων τι χρηματοπιστωτικά, χρηματοδοτικά ας πούμε, εργαλεία θα πρέπει να δημιουργηθούν για να διατηρήσουμε το νέο νόμισμα. Το θέμα είναι να έχουμε μια θεώρηση και εδώ υπάρχουν διάφορες εκθέσεις όπου υποστήριζουν την άποψη ότι το σύστημα αυτό δεν είναι ε, βιώσιμο. Εμείς δεν λέμε ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν και ποιο, τι θα χρησιμοποιηθούν. Ε, υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Δεν, έχουμε, δεν θα εστιάσουμε μόνο στον προπολογισμό επίσης. Ε, υπάρχει δυνατότητα να εκδώσουμε, ας πούμε, ε, ομόλογα ή να χρεωθούμε, πούμε, να πάρουμε δάνειο. Ε, εξορισμού βέβαια ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ούτε ελλείμματα ούτε να πάρουμε δάνειο. υπάρχουν και άλλα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ευρωζώνη για να υπάρξει δημοσιονομική σταθερότητα στις, χώρα, στις χώρες, αλλά όλα αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω και πρέπει να έχουμε την πλήρη εικόνα για τα δημοσιονομικά και τα μακροοικονομικά εργαλεία ποια είναι και Ποιο είναι ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη, που είναι ένα από τα εργαλεία για να χρηματοδοτούμε συγκεκριμένε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι ψηφίδε σε αυτό το πλαίσιο και κάποια θα δημιουργηθούν στο μέλλον ή θα αλλάξουν σχέση μεταξύ τους. Ο κύριος Μπρόκμαν έθεσε σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και έκανε και προτάσεις. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Αλλά όταν μιλάμε για ευελιξία σε αντιδιαστολή με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να πάμε από το ένα άκρο στο, στο άλλο. Η ιδέα του εφταϊτού πλαισίου είναι να, να υπάρχει μια συνέχεια στις μακροπρόθεσμες πολιτικές. Συνοχή, γεωργία, πέστε ό,τι θέλετε. Τα μεγάλα, οι μεγάλοι πυλώνες του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Εάν το κάνετε ετήσιο τον προπολογισμό, τότε θα υπάρχουν αβεβαιότητε ε, ή θα αυξηθούν οι αβεβαιοτητε προφανω είναι δυνατόν και είναι εφικτό να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη, να βρούμε μεγαλύτερη ευελιξία, παράλληλα όμως να υπάρχει μια προβλεψιμότητα στα δημοσιονομικά της Ένωσης. Και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί εν ώψη του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μου άρεσε το παράδειγμα του Λαμασούρ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και γιατί κοστίζει παραπάνω και γιατί δεν μειώνεται το κόστος ε, δεν μειώνει το κόστο που βαραίνει τι διπλωματικέ υπηρεσίε των κρατών μελών. Εγώ ξέρω τη διπλωματική υπηρεσία τη δική μου χώρα. Δεν ξέρω καμία χώρα η οποία θα παρτιθεί από τη δική τη διπλωματία. Παράλληλα όμω η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη ε, διευθύνεται και από διπλωμάτε. Τα μέλη του Κορεπέρ, έτσι, λέει ο πρόεδρο. Αλλά είναι κάτι, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, λέει ο κ. Και ε, αρνείται να το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, τι προξενικέ υπηρεσίε. Ε, μοιραζόμαστε τι υπηρεσίε, έχουμε ένα κοινό σύστημα θεωρήσεων, όλα υπάρχουν και όμω η ενιαία υπηρεσία λέει Α, όχι, εμεί δεν θέλουμε προξενικέ υπηρεσίε, κάντε τα εσεί. Εσεί, τα δικά σα προξενία. Χαχαχα. Αυτό είναι ένα α, θέμα που θα μπορούσε κάπω να επιληθεί. Να, να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προξενικέ υπηρεσίε δηλαδή, ούτω ώστε να μην διασπαθίζουμε πόρου, α πούμε, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με επιπλέον πάντα σε εθνικό επίπεδο. Πολλέ πολλές ε, και καλές ερωτήσεις έκανε ο κύριος Τεπρέ. Αν ας πούμε ε, τα πρόστιμα ε, για θέματα ανταγωνισμού θα πρέπει να πηγαίνουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή όχι, είναι ευαίσθητο θέμα, θα πρέπει να συζητηθεί και σημαντικό βέβαια. Ποια είναι η βάση για τη συνένεση. 50% σπίδιων πόρων, ας πούμε. Που θα απορρέει από ένα καλάθι πιθανών πόρων. Το 50% ήδη πόροι. Όλα αυτά προσιτηθούν. Και δεν θα πρέπει να τα αναβάλουμε. Γιατί η Κομισιόν φέτος ξεκινά, ξεκίνησε μια προσπάθεια και θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα στο τέλος. Ε, και είναι το σχέδιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα είναι η στιγμή λοιπόν να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Μελέτες, προσωμιώσεις, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι. Και να βρούμε μια καλή λύση στο τέλος του 17. Πρόεδρε, εσείς απαντήσατε στις παρατηρήσεις που ακούσαμε για την ευελιξία από τη μία προβλεψιμότητα από την άλλη του προπολογισμού. Να προσθέσω και εγώ κάτι. Πέρα από τις πληρωμές και τις διαφορές ανάμεσα στις πληρωμές και στις υποχρεώσεις, ε, συνέβη κάτι αντίστοιχο το 2013 στη Γαλλία. Η Γαλλία, θυμάμαι, έπρεπε να πληρώσει 2 δισεκατομμύρια. Και αυτό ε, δημιούργησε τον κίνδυνο για τη Γαλλία να μπει στο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δηλαδή να τιμωρηθεί γιατί το έλλειμμά τη θα αυξανόταν πολύ. Και το έλλειμμά τη αυξανόταν πολύ γιατί η Γαλλία έπρεπε να πληρώσει ε, τη συνδρομή τη στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που ήταν 2 δι. Πρέπει να συντονιστούμε λιγάκι. Δηλαδή το, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι συνεισφορέ στον προπολογισμό πρέπει να τα, να τα συνδυάσουμε καλύτερα. Δεν είναι μόνο εδώ το θέμα των ε, πιστώσεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών, το θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει, ή μάλλον συχνά τα κράτη-μέλη δεν δίνουν τη δυνατότητα στην Κομισιόν να διαχειριστεί τα οικονομικά. Κάτι πρέπει να αλλάξει, κατά την άποψή μου. κοιτάξτε τη διαδικασία. Ποιο είναι το νούμερο του γαλλικού προπολογισμού. Δηλαδή, τι, ποσό πρέπει να συμφέρει η Γαλλία στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η Κομισιόν έχει προβλέψει για τον επόμενο έτος. Οι Υπουργοί Οικονομικών συνήθω λένε «Α, η Κομισιόν μας ζητάει πάρα πολλά. Να μειώσουμε το ποσό». Πώς μειώνουμε, κανένα δεν ξέρει. Η Κομισιόν θα πρέπει να ξέρει τι ανάγκε έχει την επόμενη χρονιά. Οι υπουργοί όμω οικονομικών πάντα αποφασίζουν να δώσουν λιγότερα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και τελικά, όταν υπάρχουν ε, ε, πιστώσει υποχρεώσεων που θα πρέπει να πληρωθούν, ε, τιμολόγια που πρέπει να πληρωθούν, υπάρχουν επιπρόσθετε δαπάνε ε, κατά τη διάρκεια του έτου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούν οι εθνικοί προπολογισμοί. Υπάρχει διαδικασία δηλαδή συντονισμού των εθνικών προπολογισμών με του με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και αυτό ο συντονισμό είναι πολύ κακό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Πρόεδρε. Νομίζω ότι απάντησα στι περισσότερε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στρέφομαι προς τις κυρίες Άντολφ και Νερούτοβα. Πολύ ενδιαφέρον. ήταν και πολύ διαφωτιστικές ε, οι ομιλίε τους. Ρωτώ λοιπόν αν έχουν και αυτές σχόλια. Ευχαριστώ. Αν δούμε λιγάκι το τι μπορεί να κάνει ο ενωσιακός προπολογισμό και το τι έχει ήδη συμβάλει ε, στο να δώσει κάποια εξουσία στους πολίτες, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να δούμε λιγάκι και το θέμα των εσόδων. Και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία μας. Αν δούμε λιγάκι το μεγάλο χάσμα επενδύσεων που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη και ε, κατ' ουσίαν προκύπτει από τις τρευλώσεις της αγοράς που υπάρχουν. Νομίζω αναφερθήκατε και στα κριτήρια της βιωσιμότητας. Ε, αν τα δούμε όλα αυτά, ε, τότε θα καταλήξουμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι πρέπει να παραμείνει ως η πλέον ανταγωνιστική οικονομία. Και αυτό που σας λέω είναι απλά να δείτε λιγάκι τη θετική πλευρά των πράσινων ιδίων πόρων. Ε, ξέρω ότι η δουλειά σας είναι πολύ σκληρή. Ε, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να μιλάει κανείς για τον ενουσιακό προπλογισμό μέσα σε μια περιραίους ατμόσφαιρα Brexit. Αλλά εγώ ε, θέλησα να βοηθήσω και σας εύχομαι καλή τύχη. Η κυρία Νερούντοβα, παρακαλώ. Και εγώ περίπου τα ίδια έχω να σχολιάσω με την έννοια ότι κατά την άποψή μου ε, θα πρέπει να σας απασχολεί να κλείσει αυτό το χάσμα βιωσιμότητας για να προκύψει μια διασύνδεση ανάμεσα στις ε, ενωσιακές στρατηγικές και τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Τι? Τίποτα. Α, ε, τώρα, όσον ε, ε, αφορά την έκθεση Μόντι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Να, να ευχαριστήσω τους κυρίους Λαμασούρ και Κάρφιν, τον Επίτροπο Έτιγκερ και τις κυρίες Άντολφ και Νέρντοβα. Να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί και εγώ από την ευρία συνένεση που κατέδειξε η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε αν και όλοι αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε, κατά κάποιο τρόπο στο τέλος του δημοσιονομικού κύκλου και ότι ο κοινοτικό προπολογισμό εξαιτία των περιορισμών του έχει φτάσει στα όρια ε, ενός αντρίκελου προϋπολογισμού. Έχουμε ένα επτατές πλαίσιο απόλυτα άκαμπτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αίσθηση ότι έχει πάθει ημιπληγία, γιατί συζητά μόνο τις δαπάνες και όχι τα έσοδα και αναπόκειται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να βρουν ρυθμίσεις, διευθετήσεις, επιστροφές, μειώσεις, ε, να προβλέψουν ε, τις, ε, τους έκτακτους πόρους που θα προέλθουν από κάποια πρόστιμα. Πολύ λοιπόν λεπτή η κατάσταση και ειδικά όταν δεν υπάρχει ελαστικότητα σε απροσδόκητες ή έκτακτες καταστάσεις είμαστε υποχρεωμένοι να πολλαπλασιάσουμε τους δημοσιονομικούς δορυφόρους, τα χρηματοοικονομικά μέσα, κάτι που διαφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης για την ε, σταθερότητα, για την Ευρωζώνη, που δεν ελέγχεται ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το τυφλό σημείο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οπότε έχουμε έναν προπολογισμό που είναι ανεξήγητος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα συνεχίσει λοιπόν η Ευρώπη να γυρίζει την πλάτη στους Ευρωπαίους και να μην τους μιλάει. Όχι βέβαια, γιατί όταν εσκύπτει μια κρίση όλοι διαρωτώνται. Και η Ευρώπη τι κάνει, πού είναι. Και όταν μια χώρα οργανώνει ένα δημοψήφισμα για να παραμείνει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει κανείς την παραμονή στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι αρκετά πιστική ώστε να μην αποφασίσει η πλειοψηφία την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι ο προπολογισμό είναι η έκφραση τη πολιτική βούληση. Τι θέλουμε να πραγματοποιήσουμε από κοινού. Και τώρα προσπαθούμε με τον προπολογισμό ε, να, ε, να τραβήξουμε κάποια κονδύλια από εδώ και από εκεί και το Συμβούλιο κάνει το, παίζει το ρόλο του καλού λέγοντας «Α, κατάφερε να μειώσω τις δαπάνες της Ευρώπης», κάτι που δεν είναι ε, και πολύ θετικό για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατάλαβα όμως από τα σχόλιά σας ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χωρών, αύριο των 27. Γιατί η Ευρωζώνη εφαρμόζει μια πολύ ειδική αλληλεγγύη και όταν έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας που είναι ένα είδος Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, ε, η διαμόρφωση του κεφαλαίου δεν γίνεται από 28 χώρες μέλη, αλλά από τις χώρες της Ευρωζώνης. Και όταν έχουμε κεφάλαιο 60 δισεκατομμύρια, εσείς οι βουλευτές θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτά τα κονδύλια στον προπολογισμό. Το ίδιο ισχύει όταν θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας να προσφύγει σε δανεισμό. Τότε τα μέλη της Ευρωζώνης εγγυώνται την έκδοση ε, των ομολόγων των αξιογράφων. Επίσης, ε, ε, είπαμε να μειώσουμε τους διορθωτικούς μηχανισμούς, της μειώσεις και τις επιστροφές, που είναι πραγματικά διαφανής διαδικασία και ουσιαστικά είναι η παραχώρηση που έκανε το Συμβούλιο για να πιέσει μια χώρα να δεχτεί κάτι. Και γίνεται μια πλειοδοσία και καταφέρει μια χώρα να πετύχει μείωση και επιστροφή. Όλα αυτά είναι ε, ανεξήγητα αδικαιολόγητα και σίγουρα δεν συνάδουν με τη δημοκρατική νομοποίηση. Σε ό,τι αφορά του ιδίου πόρου, θέλουμε περισσότερου ιδίου πόρου ώστε να αποφεύγουμε να ζητούμε συνδρομέ συνεχώ από τα κράτη-μέλη και νέοι ίδιοι πόροι δεν σημαίνει κατά ανάγκη συμπληρωματικοί πόροι. Γιατί αν ο ενωσιακό προπολογισμό είχε ιδίου πόρου, είτε από τέλη που θα δίνεται από δικαιούχου ε, υπηρεσιών ή για θεωρήσεις ή για εισόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θεσπίσουμε φόρο για τον άνθρακα ή άλλους ειδικού φόρους που θα τροφοδοτούν άμεσα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τότε θα έχουμε αύξηση των υποχρεωτικών ε, ε, εισφορών, οπότε θα πρέπει να ελαφρύνουμε μια άλλη πλευρά, να μειώσουμε δηλαδή αντίστοιχα τους φόρους που, που συλλέγονται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Και διορθώστε με κύριε Ντεπρέ αν κάνω λάθος. Δηλαδή, ήδη η πόρη, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει συμπληρωματική πόρη, επιπλέον πόρη. Επίσης, τα μερίσματα που δίνει η πορη παραλαμβανω Κεντρική Τράπεζα στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, που επίσης ε, δίνουν μερίσματα στον εθνικό προϋπολογισμό, ε, τα μερίσματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί δεν πηγαίνουν κατευθείαν στον ενωσιακό προϋπολογισμό και σε αντιστάθμισμα τα κράτη-μέλη που έχουν λιγότερους πόρους να μειώνουν αντίστοιχα τη συμβολή τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και το πλεονέκτημα που θα έχουν ήδη οι πόροι που θα πηγαίνουν κατευθείαν στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, στον ενωσιακό προϋπολογισμό, είναι ότι θα ε, ε, ξεφεύγουμε από αυτό το, την δίκαιη επιστροφή που είναι προσφυλής ακόμη σε πολλές χώρες. Επίσης, ε, το ενδιαφέρον της έκθεσης είναι ότι ε, δημιουργεί μια αντιστοιχία μεταξύ τμήματος εσόδων με τμήμα δαπανών. Δαπανών που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, που είναι περιβάλλον, ενέργεια και άλλοι τομείς της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, λέμε ότι θα πρέπει να επιχειρήσουμε να καταρτήσουμε ένα προπολογισμό που θα μιλάει, θα αγγίζει τους Ευρωπαίους και θα αντιλαμβάνονται πώς γίνεται η διαχείρισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως προς την ευελιξία, την ελαστικότητα, το είπε ο κ. Ράκμαν, είναι δυνατόν ένα τεστ πλαίσιο να έχει ελαστικότητα? Πολύ δύσκολο. Ιδιαίτερα όταν 75 με 80% του προπολογισμού επιστρέφει στα κράτη-μέλη με τη μορφή κονδυλίων της κοινή γεωργικής πολιτικής, είτε διαρθρωτικών κονδυλίων, είτε κονδυλίων αλληλεγγύης. Και όταν μιλούμε για αλληλεγγύη, μήπως θα μπορούσαμε να πλουστεύσουμε κάπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα που καθιστούν ε, την οικειοποίηση τους πολύ δύσκολη, δεν γίνεται, δεν γίνεται κτήμα τους από τους Ευρωπαίους. Και επίση τα πρώτα χρόνια της, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ουσιαστικά δεν κάνουμε δαπάνε. Γιατί πρώτα θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην περιπλοκότητα των νέων προγραμμάτων. Κάτι που επίση θεωρώ σημαντικό είναι το γεγονό ότι οι Ευρωπαίοι, τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια συμφωνούν να συμπεριλάβουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό αυτό που χρειάζεται. Τι θέλουμε όμως να κάνουμε με την Ευρώπη. Μας τα ανέπτυξε διεξοδικά ο Αλάλα Μασούρ. Δεν έχουμε κάποιες αρμοδιότητες ε, κυριαρχικότητες που είναι δύσκολο να ασκηθούν σε εθνικό επίπεδο και θα είχαμε συμφέρον να τις ε, μεταφέρουμε, να τις μεταβιβάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση και το κύριο ζήτημα και γι' αυτό θα πρέπει να το φέρουμε στη δημόσια συζήτηση στα κράτη-μέλη. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε πολύ πιο στενές σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα και δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν δεν έχουμε τη συμφωνία ε, σε εθνικό επίπεδο και δεν υπάρχει αυτή η οικειοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και θέλω να έχουμε πιο τακτικές επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια με συνεδριάσεις που θα έχουν κανονική σε διάταξη, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, και ίσως και με ψηφίσματα κοινά. Γιατί όχι, γιατί να μην έχουμε κοινά ψηφίσματα των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό, που θα γίνονται αντικείμενο συζήτηση στη συνέχεια και εδώ και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμότατα. Σκεφτήκαμε, είναι έτοιμοι οι διπλωμάτες ε, να ε, μοιραστούν κάποια, κάποιους πόρους, κάποια μέσα στις εξωτερικές ε, αντιπροσωπείες. Ναι, είναι θέμα πολιτικής βολής κύριε Κάλφιν. Και εσείς τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας, γιατί βάσεις, ε, νομικές βάσεις υπάρχουν, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε την πολιτική βούληση και το πολιτικό όραμα. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει κυρίως και εκεί και το καθήκον μας, η ευθύνη μας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Να σας ενημερώσω ότι το γεύμα θα ξεκινήσει στις 1 παρατέταρτο και όχι 1 όπως είχαμε αρχικά προβλέψει. Ραντεβού στο χώρο για χούντι μενοχήν στο κτίριο Πόλαν Ρίσπακ στο πρώτο όροφο. Ε, και στον τρίτο όροφο του κτηρίου Πόλαν Ρισπακ θα βρεθούμε από τις 3 το απόγευμα, ώστε στην αίθουσα της Ελομέλειας να συζητήσουμε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο Στήματος Εθνικής Χάραξης Πολιτικής, ανταλλαγή απόψεων για τις βέλτιστες πρακτικές. Σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση.